Prendiamo corpo. Bene, diamo inizio. Ξεκινάμε. Αυτή τη σημαντική ακρόαση. Έκθεση πρωτοβουλίας του Ζωζέ Μποβέ που προτείνει συγκεκριμένες δράσεις για να μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε τα εισοδήματα μέσα στην τροφιμική αλυσίδα και τους παραγωγούς και τους καταναλωτές που πλακώνονται στην κυριολεξία στον πόλεμο των γεωργικών τιμών. Ρύθμιση του ανταγωνισμού, καταπολέμηση της κατάχρησης των ε, μεγάλων δικτύων διανομής, ε, πρόθεση συμβολέων πωλήσεων κλπ. κλπ Μία πολύ σημαντική έκθεση που και χάρη των εμπειρογνωμόνων που τους ευχαριστούμε που ήρθανε. Ε, είναι μια έκθεση σημαντική που θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα το σύστημα λειτουργίας ε, της αλυσίδας. Ε, ευχαριστώ πολλούς εμπειρογνώμ, όλους τους εμπειρογνώμονες που ήρθανε, πολύ έρχεστε από μακριά. Σας ευχαριστώ λοιπόν εξ ονόμου της Επιτροπής μας. Η αβεβαιότητα των αγορών λόγω της αστάθειας των τιμών και η αστάθεια των σχέσεων μέσα στην αγροτροφιμική ε, αγροτροφημική αλυσίδα επιβαρύνει τους ε, γεωργούς κυρίως σε τέτοιες στιγμές ε, κρίσης. Το Κοινοβούλιο ξεκίνησε διάφορες ε, ε, πρωτοβουλίε τα τελευταία χρόνια, πιο συγκεκριμένα με μία δήλωση του Ιανουαρίου του 2008, όπου προσπαθήσαμε να ξεκαθαρίσουμε τι γίνεται με την κατάχρηση εξουσίας των σούπερ μάρκετ και την, επίσης μετά εξετάσαμε το 2009 Κατόπιν πρωτοβουλία τη Κατερίνα Μπατζαλή και σήμερα Υπουργού Γεωργία στην Ελλάδα εξετάσαμε το θέμα των τιμών και τη διαμόρφωση των τιμών από, τα σούπερ μάρκετ, κάναμε μία έκθεση για το γάλα και την κατολίσθηση των τιμών του γάλακτος. Η Κομισιόν όταν παρουσίασε την ανακοίνωσή της για τον τρόπο λειτουργίας αλυσίδας φάνηκε να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στο πρόβλημα. Δίνω το λόγο τώρα στον εισηγητή, τον Αντιπρόεδρο Ζωσέ, ε, Μποβέ που θα μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσης. Και μετά θα ξεκινήσουμε με τους εμπειρογνώμονες. Και μετά συζήτηση. Ζωζέ Μποβέ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι γύρω από αυτό το τραπέζι θα ακούσετε αυτή την έκθεση. Δεν θα σας τη διαβάσω φυσικά, αλλά θα σας την παρουσιάσω σύντομα ε, για να καταδείτε τη συζήτηση πώς έχει. Το 2009 ήταν μια καταστροφική χρονιά για τους Ευρωπαίους χωρικούς. Κατά 12% μέσο όρο έπεσε το εισόδημά τους με μεγάλες ανισότητες στην Ουγγαρία χάσανε 35% έναντι του 2008 οι αγρότες, 25% στην Ιταλία και 20% στη Γαλλία χάσανε οι αγρότες. Ποιος άλλος ε, οικονομικός τομέας ε, πλήγει τόσο από την κρίση των ε, χρηματοπιστωτικών αγορών. Κάτω από το κομπρεσέρ της, τον οδοστρωτήρα της μείωσης των τιμών, πολλοί χωρικοί χρειάστηκε να κλείσουν τις εκμεταλλεύσεις τους. Πάνω από 25.000 αγρότες στην Γαλλία ε, εξαρτώνται από τα επιδόματα ε, ελαχίστου επιβίωσης που τους δίνουν οι δήμοι και οι κοινότητες. Δεν πρόκειται λοιπόν εδώ πλέον για αναδιάρθρωση, αλλά για καταστροφή των θέσεων απασχόλησης και της δυνατότητας παραγωγής των γεωργών. 14 εκατομμύρια άτομα απασχολούνται στη Γεωργία στην Ευρώπη. Η διατήρηση αυτών των θέσεων σε μια φάση όπου περνάνε κρίση όλοι οι άλλοι εργασιακοί τομεί είναι σημαντικότατο από πολιτικής πλευράς. Από το 1999 μέχρι το 2005 η προστιθέμενη αξία της τροφιμικής αλυσίδας προς τον παραγωγό πέρασε από 31% στο 24%. Όλοι οι άλλοι τομείς ε, βελτίωσαν ε, την ε, αντίστοιχη θέση τους. Και αυτό γιατί κατάφεραν να επιβάλλουν χαμηλές τιμές, χαμηλότερες και από το κόστος παραγωγής στους γιοργούς τους, δεν τους επέτρεψαν να βαρύνουν στη διαπραγμάτευση έναντι επιχειρήσεων πολλές φορές διεθνού χαρακτήρα. Όπως το δείχνει και η ανακοίνωση της Κομισιόνα, αυτό το σοκ των γεωργών δεν είναι υπέρ των καταναλωτών. Βλέπουμε ε, στα, ο προπολογισμό των νοικοκυριών έχει αυξήσει ιδιαίτερα τις, ε, τις ε, αγορές τροφίμων. Ελάχιστα τα σούπερ μάρκετ μείωσαν τις τιμές. Το 2009 τον Οκτώβριο όταν οι γαλακτοπαραγωγή χύνανε το γάλα του στα χωράφια, η μεγαλύτερη αλυσίδα διανομής στην Ευρώπη χαιρότανε που έβγαλε 10 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα καθαρό κέρδος λόγω των χαμηλών γεωργικών τιμών. Είναι, πολύ πιο, είναι δύσκολο να είναι κανείς αφέστερος. Η έκθεση της Κομισιόν αφορά στη σχέση μεταξύ γεωργών, πολυεθνικών εταιριών, διανομή, που εκφράζεται κυρίως από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και τους τελικούς καταναλωτές. Αυτή η αλυσίδα δεν καλύπτει σε τίποτα την πραγματικότητα. Κατά τις εβδομάδες προετοιμασίας της εκθεσής μου συνάντησα τους πρωταγωνιστές αυτής της αλυσίδας που μου ε, υπέβαλαν το αίτημα και οι ανταλλαγές που είχαμε μου παρουσίασαν πραγματικά τις ε, κόντρες, τις μεγάλες κόντρες που υπάρχουν μεταξύ παραγωγών και μεγάλων κέντρων διανομής. Δεν μπορούν δηλαδή να προχωρήσουν σε ισότιμες διαπραγματεύσεις. και τα κέντρα διανομής ε, έδειξαν ιδιαίτερη μυστικοπάθεια στο να πούνε ποιο είναι το περιθώριο το κέρδους τους. Η διαφάνεια των τιμών είναι αναγκαιότητα πλέον. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθούν διεπαγγελματικοί κλάδοι οι οποίοι να ενώνουν όλους τους κρίκους της αλυσίδας από το χωράφι στο πιάτο για να μπορέσουμε να δούμε πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Γιατί το σιτάρι είναι μόνο το 5% στην τιμή ενός καρβελιού ψωμί και ένα κιλό μήλα το οποίο το πληρώνουν 10 σέντ στον παραγωγό, το πληρώνει ο καταναλωτής 2 ευρώ. Πρέπει να δούμε ποιο είναι το καθαρό περιθώριο των εκμεταλλεύσεων οι οποίες βρίσκονται ε, παγιδευμένες ε, μεταξύ της ε, βιομηχανίας υποδομών, δηλαδή γεωργικών μηχανών, σπόρων κλπ. και της μεγάλης διανομής. Να σας δώσω δύο παραδείγματα. Τα, τα πέντε βασικά σούπερ μάρκετ στη Σουηδία εμπορευματοποιούνται το 80% των τροφίμων, στη Γαλλία 70%. Αυτή η συγκέντρωση οδηγεί σε, σε έναν πόλεμο των τιμών που οδηγεί στην αναζήτηση των φτηνότερων γεωργικών προϊόντων της εντατικής γεωργίας η οποία δεν αναλαμβάνει το πραγματικό της κόστος, δηλαδή μολύνει νερό και έδαφος ξοδεύει ενέργεια, εκπέμπει αέρια θερμοκηπίου και δεν τα λέει όλα. Και ομοιομορφοποιεί τις ε, τροφιμικές ε, συνήθειες. Το περιβάλλον, ε, η παραγωγή, ο καταναλωτής και ο φορολογούμενος είναι οι μεγάλοι χαμένοι αυτού του, αυτού του αγώνα τρεξίματος, αυτής κούρσας. τα μικρά μπακάλικα στην, ε, στην Ήπεθρο ε, ή στην, ε, σε δύσκολες γειτονιές της πόλης πλήττονται από όλη αυτή την ιστορία επίσης. Ο κόσμος για να κάνει τα ψώνια του σήμερα πρέπει να πηγαίνει συνεχώς περισσότερο με αυτοκίνητο. Στην τροφιμική αλυσίδα οι καταχρήσεις και οι δεσπόσουσες θέσεις είναι τεράστιες, αλλά δύσκολο να αποδειχθούν. Οι γεωργοί και οι Ε που είναι και τα θύματα διστάζουν συχνά στο να υπερασπίσουν τα δικαιώματά τους και αυτό γιατί φοβούνται μη χειροτερεύσει κατάσταση. Ζητώ λοιπόν από την Κομισιόν να συντάξει μία έκθεση για όλες αυτές τις καταχρήσεις και πιο συγκεκριμένα στις καταχρήσεις εκείνες οι οποίες ε, έχουν να κάνουν με την επαναχρηματοδότηση, με τις επιστροφές με την μεταπόληση με χάσιμο κλπ. Θα πρέπει να είναι αμετάκλητη η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά και να καταστήσει αυτές τις πρακτικές παράνομες, όπως κάνανε και σε ορισμένα κράτη-μέλη, Γερμανία, Ισπανία, Ιρλανδία, Γαλλία. Να πληρώνουν δηλαδή, ε, να πουλούν με απώλεια και να γκρεμίζουν την ε, ε, κάθε αρχή ανταγωνισμού. Θα πρέπει να σταματήσουν αυτές οι πρακτικές. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε πραγματικές οργανώσεις παραγωγών που θα μας επιτρέπουν να προχωρούμε σε συλλογικές διαπραγματεύσεις και να ελέγχουμε την παραγωγή για να έχουμε μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Όπως είπαμε και πριν, η ευρωπαϊκή τροφιμική Λυσίδα δεν είναι μονολυθική. Η πώληση, η απευθείας πώληση από τον παραγωγό στον καταναλωτή ε, υπάρχει ε, και γίνεται χωρίς να μολύνει το, το, το, περιβάλλον ε, και προτείνοντας δίκαιες τιμές αλλά επλήγει κυρίως από όλα τα μέτρα υγειονομικής προστασίας που ευνοούν τις μεγάλες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να ξαναδούμε όλα αυτά τα μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη την τη μικρή παραγωγή και τα μικρά κέντρα πώλησης. Ε, εμείς, ε, παραδειγματικά, η οικογενειακή κήπη, οι μπαξέδες, τα περιβόλια στη Γαλλία είναι 250.000 εκτάρια και η οικογενειακή παραγωγή ντομάτε, ντομάτας είναι το 1 τέταρτο της, εθνικής, της ετήσιας εθνικής κατανάλωσης. Σε άλλα κράτη-μέλη όπως η Ρουμανία, οι συνταξιούχοι παράγουν το 1 τρίτο των ε, τροφιμικών τους αναγκών. Αυτά τα ποσά δίνουν και μία οπτική της τροφιμικής αλυσίδας που είναι σχεδόν άγνωστη ή δεν αναφέρεται σχεδόν καθόλου το ότι υπάρχουν στην Ευρώπη 40 εκατομμύρια άτομα που εξαρτώνται από τις τράπεζες τροφίμων για να φάνε είναι αποτυχία. Μία από τις βασικές αιτίες αποτυχίας της ΚΑΠ. 80 εκατομμύρια άτομα έχουν δυσκολία να ταΐσουν την οικογένειά τους η μείωση των τιμών προς τους χωρικούς ε, δεν επέτρεψε να αλλάξει η τάση. Η ανεργία, η μείωση εισοδήματος, η χαμηλή μισθή, οι γελίες συντάξεις είναι ο βασικός λόγος δυσκολιών των συμπολιτών μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξήγαγε το 2009 23 εκατομμύρια τόνου στάρι και ξεπούλησε τα πλεονάσματα σε γάλα και σε κρέας στις παγκόσμιες αγορές. Αυτό δεν έχει να κάνει λοιπόν με έλλειμμα παραγωγής και παραγωγικότητας, αλλά με κοινωνική αηδία σε μία άνηση κατανομή εισοδημάτων στην Ευρώπη για να μην μπορέσουν, για, για να μην ενισχύσουμε εμείς όλες τις καμπάνιες φιλανθρωπίας αλλά να ενισχύσουμε την αξιοπρέπεια θα πρέπει η Ευρώπη να παλέψει για την αυτάρκεια. Θα πρέπει να δοθεί κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα και αυτά να θεωρούνται προτεραιότητες. Το 2007 όταν οι γεωργικές οι πρώτες ύλες είχαν φτάσει στα ύψη, ορισμένες ευρωπαϊκές τράπεζες άρχισαν να κυνηγάνε τους, τους ε, πελάτες τους στο τηλέφωνο για να αρχίσουν να επενδύουν στα παράγωγα κεφάλαια, στα κερδοσκοπικά κεφάλαια βραχυπρόθεσμα τα οποία οδήγησαν καθοδήγησαν και την ε, τάση ε, των γεωργικών προϊόντων. Και αυτού του είδους η πολιτική είναι και η βασική αιτία για, όλες, ε, για όλα τα ξεσπάσματα κινητοποίησεων και στάσεων στις χώρες του Νότου. Θα πρέπει τα, οι γεωργικές πρώτες ύλες να μην επηρεάζονται από το γενικό χρηματιστήριο. Να μην είναι και οι γεωργικές πρώτες ύλες κερδοσκοπικά ε, κερδοσκοπικό αντικείμενο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κοιτάξει να θέσει διεθνή μέσα ρύθμισης, να το δει και με τους εταίρους της τι μέτρα κατεπήγοντα πρέπει να ληφθούν, ούτω ώστε η χρηματοπιστωτική σπέκουλα να μην καταστρέφει τους ε, γεωργούς, ε, τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και να αποστεθαροποιεί την ΚΑΠ η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ γύρω από την οποία εργαζόμαστε θα καταφέρει αν μπορέσουμε εμείς να εξισορροπήσουμε το συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ των διαφόρων πρωταγωνιστών της αλυσίδας να, να ρυθμίσει την προσφορά και να καταπολεμήσει την κερδοσκοπία για να μπορέσουμε εμείς να, να μπορέσουν να υποφεληθούν οι συμπολίτε μας από ποιοτικά καλά γεωργικά προϊόντα. Εισόδημα λοιπόν δίκαιο για τους Ευρωπαίους Γιωργούς, προστασία του περιβάλλοντος και αρμονικό οικονομικό-κοινωνικό περιβάλλον στην επικράτειά μας. Αυτός είναι ο στόχος της έκθεσής μου. Να συμμετέχουμε όπως το έκανε και ο κύριος Λάιον για την ΚΑΠ στην οικοδόμηση αυτής της νέας ΚΑΠ που θέλουμε όπως την επιθυμούμε μετά το 2013 ώστε ο καθένας από εμά να ξαναβρει την αξιοπρέπειά του και να μπορεί να ζει από το εισόδημά του στο χωριό. Ευχαριστώ τον Ζωζέ Μποφέ. Σας ευχαριστώ και για το πάθος με το οποίο παρουσιάσαστε στην την εκθεσή σας και τώρα να δώσουμε το λόγο στους εμπειρογνώμονες. Έχουμε επτά προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες, έτσι λοιπόν θα ήθελα να απευθύνω μια έκκληση να περιοριστείτε στα 10 λεπτά για το χρόνο ομίλια σας. Σας ξεκινήσουμε τον κύριο Όλιβερ Ντεσούτερ, ο οποίος είναι ειδικό εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για το δικαίωμα στη διατροφή. Κύριε Ντεσούτερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η εντολή που μου έδωσε το Συμβούλιο των Δικαιωμάτων Ανθρώπου είναι να εργαστώ επί της ε, πρόθεση του δικαιώματο τη διατροφή ε, στον κόσμο και μπορώ να σας πω ότι από τα εκατομμύρια ανθρώπων ε, που πεινούν σήμερα πάνω από τα δύο τρίτα ε, παράγουν την τροφή τους. Έχουμε 650-700 εκατομμύρια ανθρώπους που πεινούν και έναν αριθμό παραγωγών και στις αναπτυσσόμενες χώρες όπως και στην Ευρώπη. Βλέπουμε ότι οι τιμέ συνεχίζουν να ανεβαίνουν ανεβαίνουν στα τρόφιμα ενώ ε, οι τιμέ στον παραγωγό συνεχίζουν να μειώνονται. Βλέπουμε εδώ ότι έχουμε ιστορικού παραγωγού οι οποίοι εδώ και 30 χρόνια έχουν τεθεί στο περιθώριο από την βιομηχανική παραγωγή και δεν μπόρεσαν να στηρίξουν την παραγωγή του. Πρόκειται για μικρού γεωργού που σήμερα ζουν από μια γεωργία επιβίωση, που του επιτρέπει μόλι να επιβιώσει και κατόπιν έχουμε 200-200 εκατομμύρια άτομα που πεινούν και πρόκειται για άτομα που εργάζονται σε μεγάλες φοιτίες, είναι εργάτες στον τομέα της γεωργίας ε, και ε, βιώνουν έναν ανταγωνισμό σε διεθνές επίπεδο με την απελευθέρωση του εμπορίου των ε, αγροτικών προϊόντων και αυτό μας οδήγησε στην μείωση των μισθών αυτών των εργαζομένων και μάλιστα σήμερα σήμερα δεν χαίρουν ε, και νομική προστασία. Η μεταμόρφωση τη Γεωργία σε παγκοσμίο επίπεδο οδήγησε σε αυτή την καταστροφική κατάσταση που έχουμε σήμερα. Δηλαδή ένα δισεκατομμύριο ανθρώπου ε, να υποφερούν από την πείνα και αυτό αποτελεί αποτέλεσμα πολιτικών που ευνόησαν ένα είδο Γεωργία δηλαδή την γεωργία μεγάλης κλίμακας, ε, ιδιαίτερα βιομηχανοποιημένη που δεν είναι ούτε πλέον η πιο παραγωγική ένα εκτάριο, αλλά ούτε και η πιο αηφόρος από κοινωνική και περιβαλλοντική σκοπιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα έχω την ευκαιρία να απευθυνθώ εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να αναπτύξω εις βάθος το σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ της ρύθμισης της διατροφικής αλυσίδας στην Ευρώπη και του επιστημιστικού τομέα, γεωπιστημιστικού τομέα σε εθνικό σε διεθνέ επίπεδο, με συγχωρείτε. Πρέπει εδώ να δράξουμε την ευκαιρία που μα προσφέρει η ανακοίνωση τη Κομισιόν για να εξετάσουμε την ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εναντί τη ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή τη ε, αλυσίδα εφοδιασμού των τρεφίμων. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε τέσσερα σημεία. Έχετε στη διάθεσή σας ένα κείμενο όπου αναπτύσσονται ε, πολύ λεπτομερέστερα τα στοιχεία που θα σας αναφέρω προφορικά. Καταρχήν, ε, έχουμε το θέμα της συγκέντρωσης στο γεωπιτιστικό τομέα. Αυτή η συγκέντρωση έχει συνέπειες καταρχήν οδηγεί στο εξή. Μέσα στον ίδιο τον γεωπιστικό τομέα, στην αλυσίδα, μία ε, μικρή αναλογία τη προστιθέμενη αξία, δηλαδή αυτό που πληρώνει τελικά ο τελικό καταναλωτή, σε ένα πολύ μικρό κομμάτι να πηγαίνει στο γεωργό, στον παραγωγό και στι ε, παραγωγικέ χώρε. Έχουμε πολλά αριθμητικά στοιχεία που μας δείχνουν πώς αυτή η αναλογία ε, του εισοδήματος συνεχίζει να μειώνεται για τον παραγωγό. Ε, πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτή την υπερβολική συγκέντρωση και κατά τις δεσπόζουσες ε, θέσεις που σχετίζονται με αυτά. Υπάρχουν όμως ε, προβλήματα στο σημερινό σύστημα. Καταρχήν το δικαίωμα στον ανταγωνισμό και στην δημιουργία κέρδους, όχι για τον παραγωγό το δικαίωμα στον ανταγωνισμό μέχρι σήμερα έχει χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τον καταναλωτή έτσι ώστε ο καταναλωτής να μην πληρώνει υπερβολικά ακριβά τα προϊόντα και πρέπει να σκεφτούμε την δυνατότητα να ξανασχεδιάσουμε την πολιτική ανταγωνισμού, να δούμε ποιο είναι το ισχυρό νομικό καθεστώς για το δικαίωμα του ανταγωνισμού, για να δούμε αν ο πολιτής ε, θα πρέπει να είναι προστατευμένο έναντι της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης ε, που πολλέ φορέ χαρακτηρίζει τη θέση του αγοραστή. Η δεύτερη δυσκολία είναι ότι στην παγκόσμια ε, αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων που σχετίζει τον παραγωγό του Νότου με τον καταναλωτή του Βορρά, πολύ συχνά υπάρχουν προβλήματα εξοδαφικότητας και το δικαίω του ανταγωνισμού δεν καλύπτει το ζήτημα αυτό. Οι ίδιες αναπτυσσόμενες χώρες δεν έχουν ε, δικαίωμα στον ανταγωνισμό και αν υπάρχει, εφαρμόζεται ελάχιστα. Πώ μπορούμε να εξηγήσουμε λόγω χάρη, παραδείγματο χάρη, εκ του ε, να ε, έρθει, παραδείγματο χάρη, σε αντίθεση με την εταιρεία που εκμεταλλεύεται τι φοιτίε κακάο. Επίσης, ε, σε ό,τι αφορά τώρα το δίκαιο του ανταγωνισμού που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, πολλές φορές ε, είναι δύσκολο να εφαρμοστεί εξωεδαφικά, εκτός αν θίγεται η εσωτερική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή αν θίγονται τα δικαιώματα των Ευρωπαίων καταναλωτών. Πιστεύω ε, ότι είναι καλή η πρόταση που έγινε από τον κύριο Μποβέ να εξηγήσουμε αν ε, το δικαίωμα στον ανταγωνισμό θα πρέπει να βελτιωθεί για να δούμε ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα που τίθεται στο γεωπιστικό τομέα καθώς αυτά τίθεται σε ένα όλο ένα και πιο παγκόσμιο επίπεδο και όχι συγκεντρώσεις δεν περιορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια άλλη συνέπεια της συγκέντρωσης είναι ότι αγοραστές ε, στην αλυσίδα εφοδιασμού συχνά εφαρμόζουν καταχρηστικέ πολιτικές. Σε μια έκθεση που υπέβαλα ε, τον περασμένο Μάρτιο στο Συμβούλιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, αναφέρθηκα στα προβλήματα που ανέφερε και ο Ζωζέ και νομίζω ότι ίσως ε, ε, πιο συστηματική προσέγγιση είχαμε σε αυτό τον κώδικα πρακτικών που ανέπτυξε το Ηνωμένο Βασίλειο και ανέφερε όλες τις πρακτικές που θα πρέπει να απαγορεύονται από την πλευρά των αγοραστών και ουσιαστικά τίθεται σε εφαρμογή γιατί οι αγοραστές βρίσκονται σε δεσπόζουσα θέση. Νομίζω ότι υπάρχουν ε, περιπτώσεις όπου η ισορροπία της ε, σχέσης ε, ισχύων είναι τέτοια μεταξύ καταναλωτή και παραγωγού όπου θα αιτιολογούταν μια νομική παρέμβαση. Δηλαδή πολλές φορές οι παραγωγοί βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, δεν μπορούν να έρθουν σε διαπραγμάτευση με τους αγοραστές δεν έχουν εναλλακτική αν θέλουν να διοχετεύσουν τα προϊόντα τους σε απομακρυσμένες αγορές και δεν έχουν εναλλακτική παρά να περάσουν από αυτούς τους αγοραστές που κατέχουν τη δεσπόζουσα θέση στην ελισίδα. Εγώ, ε, ένας, θα έλεγα ότι ένας από τους τρόπους να ενισχύσουμε την, ε, το δικαίωμά τους, την εξουσία τους στη διαπραγμάτευση είναι να ενισχύσουμε την τοπική αγορά, δηλαδή την ε, μικρή αλυσίδα σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να έχουν Υπάρχουν ε, και άλλους τρόπους να διοχετεύσουν τα προϊόντα τους. Ένα δεύτερο σημείο αφορά την διάδοση των ε, ιδιωτικών προτύπων στο επιστημιστικό τομέα. Αυτά τα πρότυπα ενίοτε αφορούν κοινωνικές ή περιβαλλοντικές ρήτρες που επιβάλλονται στο παραγωγό, αλλά πολύ πιο συχνά στην πραγματικότητα αφορούν σε ζητήματα υγείας των καταναλωτών και επιστημιστικής ασφάλειας. Αυτές οι ρήτρε όταν επιβάλλονται στους μικρούς παραγωγούς ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν σεβαστές από αυτούς και αποτελούν ε, ένα είδος διχοτόμησης ε, του τομέα. Δηλαδή, οι μεγάλοι παραγωγοί πολύ πιο εύκολα μπορούν να σεβαστούν τα πρότυπα αυτά σε σχέση με τους μικρούς παραγωγούς και αναφέρομαι κυρίως στους μικρούς παραγωγούς σε αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίοι πολύ συχνά αδυνατούν να σεβαστούν τα πρότυπα αυτά και επομένως δεν μπορούν μπορούν να ε, διοχετεύσουν τα προϊόντα τους ε, στην αλυσίδα σε παγκόσμιο επίπεδο. Όταν ε, οι διανομή οι αγοραστές επιβάλλουν τέτοια πρότυπα στους προμηθευτές τους, θα έπρεπε να μετρήσουν τον αντίκτυπο των πρότυπων αυτών στους πλέον φτωχούς παραγωγούς, στους πιο μικρούς παραγωγούς. Θα έπρεπε να υποστηρίξουν αυτούς τους παραγωγούς προκειμένου να τους επιτρέψουν να σεβαστούν τα πρότυπα αυτά. Και θα έπρεπε επίσης όχι απλώς ε, να ε, προβαίνουν σε εποπτεία του σεβασμού, αλλά να διευκολύνουν και το σεβασμό και να στηρίζουν και οικονομικά αυτού του παραγωγού προκειμένου και αυτοί να μπορέσουν να συμμετέχουν στην αλυσίδα παραγωγής και διανομής. Τρίτον, Νομίζω ότι ένα εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά το οποίο το υποτιμούμε, είναι οι δημοσίες προμήθειες. Σήμερα το 15% του ε, ακαθάριστου κορπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δαπανάται από ε, το δημόσιο στα τρόφιμα ε, μέσω διαγωνισμών. Νομίζω ότι σε όλα τα επίπεδα, σε επίπεδα εθνικών κυβερνήσεων, αλλά και κυρίως και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αυτές οι δημόσιες προμήθειες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με ένα πολύ πιο στοχευμένο τρόπο για να ενθαρρύνουμε μια υπεύθυνη αηφόρο γεωργία η οποία να σέβεται και το περιβάλλον και να υποστηρίξουμε έτσι το δίκαιο εμπόριο. Νομίζω ότι η οδηγια 2014 2004-18 η οποία είναι πλέον σημαντική οδηγία που υιοθετήθηκε για το θέμα των δημοσίων προμηθειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια οδηγία η οποία είναι απόλυτα συμβατή με την εισαγωγή κοινωνικών και περιβαλλοντικών ρητρών και οι ρήτρε αυτέ είναι χρήσιμε χρήσιμες ε, προκειμένου να αναπτυχθεί η διατροφική αλυσίδα με πιο εύφορο τρόπο. Τέταρτο και τελευταίο. Έχουμε το θέμα της αστάθειας ε, των τιμών ε, στις διεθνείς αγορές. Αναφέρθηκε αυτό και αναφέρθηκε και ο ρόλος των κερδοσκόπων στην αστάθεια αυτή των τιμών. Πρόκειται για μια ανησυχία πραγματική το Μάρτιο του 2008, τη στιγμή που δημιουργήθηκε αυτή η κερδοσκοπική φούσκα ε, σε ό,τι αφορά τις προθεσμιακές συναλλαγές, ε, υπήρξε ε, επένδυση 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις προθεσμιακές συναλλαγές. Δηλαδή είχαμε πολύ περισσότερα δισεκατομμύρια και δύο φορές περισσότερα από το 2005. Έτσι λοιπόν αυτό δημιούργησε ε, μία φούσκα ε, για το ρύζι, ε, το καλαμπόκι, τη σόγια και είδαμε ότι μπήκαμε σε ένα σπιράλ το οποίο αναπτύχθηκε στη συνέχεια καθώς η δημιουργία αυτών των κερδοσκοπικών φουσκών για τις προθεσμιακές συναλλαγές οδήγησε τους εμπόρους να κερδοσκοπήσουν και να επιβάλλουν περιορισμού στι εξαλλαγέ ή να αποθηκεύσουν ε, εμπορεύματα, ελπίζοντα ότι θα συνεχιζόταν η να αποθηκευσουν εμπορευματα ελπιζοντα οτι θα συνεχιζοταν η ενοδο των τιμών. Αυτό πρέπει να το ρυθμίσουμε. Η G20 δεσμεύτηκαν στο Λονδίνο τον Απρίλιο του 2009 να ρυθμίσουν τα επενδυτικά ταμεία που αποτελούν συστηματικό κίνδυνο για την οικονομία. Αυτά τα επενδυτικά κεφάλαια ε, αποτελούν συστημικό κίνδυνο για την οικονομία. Πρέπει να τα ρυθμίσουμε. Μπορεί να γίνει αυτό με διάφορους τρόπους. Προτείνω διάφορες προσεγγίσεις, εκ των οποίων ε, κάποιες συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση που υπέβαλα στον ΟΗΕ και μπορείτε να βρείτε και σχετικά στοιχεία στο σημείωμά μου. Να κλείσω κάνοντας πολύ σύντομα πέντε προτάσεις. Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να δράξει την ευκαιρία να κάνει αυτή τη συζήτηση για την διατροφική αλυσίδα στην Ευρώπη για να σκεφτεί πώς μπορεί να βελτιώσει την πολιτική ανταγωνισμού δηλαδή να εργαστεί επί των φαινομένου των συγκεντρώσεων και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν ε, είναι ανεκτό το η παραγωγή στις αναπτυσσόμενε χώρες να είναι θύματα δεσπόζουσας θέσης και να πρέπει να εκχωρούν τι οδιέ του σε τιμέ που ε, με τα του επιτρέπουν να επιβιώσουν απλώς γιατί δεν έχουν άλλη δυνατότητα παρά να περάσουν από αυτού του μεγάλους αγοραστές για να έχουν πρόσβαση στις διεθνεί αγορές. Θα πρέπει επίση να σκεφτούμε ε, πώς μέσω της ρύθμισης θα κατεπολεμήσουμε τις καταχρηστικές ε, θέσεις ε, από την πλευρά των αγοραστών. Θα πρέπει επίσης ο ιδιωτικός τομέας, οι αγοραστές να προτρινθούν να εξετάσουν τον αντίκτυπο των προτύπων που επιβάλλουν ε, για ε, τη δυνατότητα που έχουν οι πιο μικροί παραγωγοί να σεβαστούν τα πρότυπα αυτά και θα πρέπει τα πρότυπα αυτά να προσδιοριστούν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν ε, προβαίνουν στο κατακαιρματισμό του τομέα. Νομίζω επίση ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο των δημόσιων προμηθειών για να αναπτυχθεί η επιστηστική αλυσίδα με πιο βιώσιμο τρόπο και νομίζω ότι και το δίκαιο εμπόριο θα μπορούσε να ενθαρρύνει μέσω πιο συστηματική προσφυγή τα προϊόντα του δίκαιου εμπορίου να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη και την αποκεντρωμένη εξουσία νομίζω ότι πρέπει να ρυθμιστεί και η συμπεριφορά των επενδυτών στις προθεσμιακές συναλλαγές και να πω ότι ένας από τους πιο σημαντικούς αντικτύπους που οι ευρωπαϊκές πολιτικές ε, είχαν στο παρελθόν ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες και στους παραγωγούς τους είναι το dumping ε, των ε, πρώτων, των γεωργικών πρώτων υλών ε, σε αυτές τις χώρες, καταστρέφοντας μια σειρά τομέων στις χώρες αυτές. Δηλαδή είδαμε πολλές φορές στις αγορές αυτές έφταναν προϊόντα τα οποία λάμβαναν ισχυρές επιδοτήσεις. Ε, έτσι λοιπόν πρέπει να κρίσουμε τον κόδωνα του κινδύνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το φαινόμενο αυτό. Πρέπει να περιορίσουμε το φαινόμενο του ντάμπινγκ και να καταργηθούν ε, οι εξαγωγικές ε, επιδοτήσεις που προκαλούν τον ντάμπινγκ αυτό και νομίζω ότι ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη μικρών αλυσίδων στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καταλήξουμε σε μια καλύτερη ρύθμιση των γεωργικών αγορών σε διεθνές επίπεδο. Σας ευχαριστώ και αν υπάρχουν είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Ντεσίτερ. Τώρα θα δώσουμε στο λόγο στον κύριο Ρότζετ Κλάρκ, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Κάρδιφ, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις άδικες πρακτικές που επιβάλλονται στους γεωργούς και θα μας μιλήσει και για το δίκαιο του ανταγωνισμού στην Ευρώπη. Έχετε το λόγο. Okay, Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μου ζητήθηκε να μιλήσω για το πώς θα πάψουν οι στρεβλώσεις ανταγωνισμού σε βάρος των γεωργών. Είμαι πανεπιστημιακός δάσκαλος στο Πανεπιστήμιο του Κάρδιφ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λόγω και του περιορισμένου χρόνου που διαθέτω, νομίζω ότι θα εγκύψω σε δύο θέματα. Ένα πιο γενικό που ήδη εφήγει σε κάποιο βαθμό και που ισχύει όχι μόνο για τους γεωργούς αλλά και για παντός είδους πρόσωπα που διαθέτουν τα προϊόντα τους, πολλούν τα προϊόντα τους και ένα άλλο πιο ε, συγκεκριμένο που έχει πιο πολύ σχέση με τους αγρότες, όχι απαραίτητα τους αγρότες ε, που παράγουν δημητριακά, αλλά και σε ορισμένες άλλες αγορές. Αρχίζω με το πρώτο λοιπόν, που όπως είπα εφήγει ήδη σε κάποιο βαθμό. Γνωρίζουμε νομίζω όλοι ότι οι αλυσίδες υπερκαταστημάτων ε, είναι εμπλεγμένες σε κάποιες ε, συμβατικές πρακτικές πρακτικές που ως αποτέλεσμα έχουν την επιβολή πρόσθετου κόστους στους πολιτές, τους πολλούν δηλαδή τα προϊόντα τους, ταυτόχρονα αυξάνουν τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν τα πρόσωπα αυτά και βέβαια αυτό πλήττει ιδιαίτερα μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι εκμεταλλεύσεις. Οι πρακτικές αυτές έχουν συζητηθεί ήδη τις οποίες ε, έχω ε, περιλάβει στη διαφάνεια αυτή που ίσως, ίσως βλέπετε, όπως για παράδειγμα καθυστερήσει στις πληρωμές, εκ των υστέρων ε, αλλαγές στους όρους προμήθειας, αν για παράδειγμα σε κάποιο έτος είχαν υψηλές πωλήσει, επίσης να πληρώνουν οι παραγωγοί για να περιληφθούν στις λίστες των υπερκαταστημάτων. Επίσης άλλα πράγματα όπως ειδικέ πληρωμές όπου ζητούν τα σούπερ μάρκετ να τους καταβληθούν ε, έξτρα πληρωμές για να ανοίξουν κάποιο ε, νέο κατάστημα ή κάτι τέτοιο. Όλα αυτά λοιπόν είναι συμβατικές πρακτικές, πρακτικές ε, εδώ στο πλαίσιο συμβάσεων, οι οποίες βέβαια είναι πρακτική των, ε, ε, ε, των σούπερ μάρκετ και ταυτόχρονα βέβαια ως αποτέλεσμα έχουν την μείωση των εισοδημάτων των πολιτών, των παραγωγών δηλαδή, και βέβαια και την αύξηση του κινδύνου τους. Αυτές οι πρακτικές είναι συνήθεις στην Ευρώπη, είναι ευρέως διαδεδομένες. Υπάρχει και μια ομάδα υψηλού επίπεδου η οποία συνήλθε και εξέτασε αλλαγές, αλλαγές που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ένα κώδικα διοντολογίας όπως υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ίδιο και η Ιρλανδία ε, καταθέτει σχετική πρόταση. Ε, με τον τρόπο αυτό μπορούν να απαγορευτούν ορισμένε πρακτικές. Φαίνεται να είναι λογικό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρξει ένα είδος κανονισμού που να μπορέσει να αποτρέψει τα σούπερ μάρκετ από του να ε, ασκούν τέτοιες πρακτικές. Υπάρχει και μια άλλη δυνατότητα. Ένα τέτοιο κώδικα διοντολογία, δηλαδή η κώδικα πρακτική, εφόσον ισχύσει, μπορεί να επιβληθεί. Ισχύει αυτό ήδη στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Να περιλάβει και έναν εξάρτητο όργανο επιβολής το οποίο έχει ονομαστεί Ombudsman στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, ε, υπάρχουν και επιχειρήματα υπέρ της επιβολής και στο ευρωπαϊκό επίπεδο με την έννοια ότι ορισμένες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου είναι πολυεθνικές και είναι δύσκολο να γνωρίζει κανείς ποιος είναι ο εθνικός οργανισμός, η εθνική αρχή η οποία θα πρέπει να ασχοληθεί, να επιληφθεί των υποθέσεων που ε, ενδεχομένως αποτελούν παραβιάσεις ενός τέτοιου κώδικα διοντολογίας ένα τέτοιο ευρωπαϊκό όργανο θα μπορούσε να επιλαμβάνεται υποθέσεων οι οποίες δεν εντάσσονται εύκολα, ας πούμε, στο νομικό πλαίσιο μιας μεμονωμένης χώρας μέλους. Αυτές είναι λοιπόν οδοί που μπορεί να εξετάσει κανείς. Έτσι λοιπόν, ένας ανεξάρτητος κώδικας πρακτικών ιδεοτολογίας για τις αλεξίδες υπερκαταστημάτων και ταυτόχρονα η μελέτη του ενδεχομένου να υπάρξει ένας ανεξάρτητος οργανισμός, ένα πρόσωπο, ένα ομπούτσμαν, ο οποίος να επιλαμβάνεται της επιβολής του ε, κώδικα αυτού. Α, αυτό λοιπόν είναι το πρώτο θέμα που επιθυμώ να θέσω στη συζήτηση. Είναι γενικής εφαρμογής σε στις διάφορες πτυχές των ε, προϊόντων που πουλούνται στα υπερκαταστήματα, γιατί δεν είναι βέβαια μόνο τα τρόφιμα, ούτε μόνο οι αγρότες οι οποίοι ε, υφίστανται τις ερισμένες συνέπειες. Και κάτι το οποίο είναι πιο συγκεκριμένα για τους αγρότες, ότι δηλαδή τα σούπερ μάρκετ και με την αγοραστική τους δύναμη έχουν προκαλέσει πρόσθετα προβλήματα στις ε, αγορές αγροτικών προϊόντων. Η οικονομική θεωρή ε, γι' αυτό, ζητώ συγγνώμη από όσους ε, τα γνωρίζετε ήδη, πάντως με δύο λόγια η θεωρία περιλαμβάνει το εξής βασικό επιχείρημα. Αυτό το χαρακτηριστικό βασίζεται στην δομή του κόστους στον κλάδο. Υπάρχουν δύο βασικά περιπτώσεις. Είτε όπου όλες ε, οι προμήθειες έχουν το ίδιο κόστος μονάδας, εκεί μπαίνει η αγοραστική δύναμη των σούπερ μάρκετ, υπάρχει και η κατάσταση ότι όπου υπάρχουν οι ίδιες καμπύλες κόστους και στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει δυνατότητα να ασκήσουν τα, τα σούπερ μάρκετ έξτρα αγοραστική δύναμη. Η άλλη δυνατότητα είναι να υπάρχουν αυξανόμενο, υπάρχει αυξανόμενο ελάχιστο κόστος με την έννοια ότι ορισμένη παραγωγή είναι πιο περιθωριακή από άλλους. Αυτό ίσως ισχύει σε ορισμένους αγροτικούς τομείς και στην περίπτωση αυτή το σημαντικό είναι όπου υπάρχουν δηλαδή διαφορετικές επιχειρήσεις με διαφορετικές μονάδες ελάχιστου κόστους είναι ότι υπάρχει κίνητρο για τους αγοραστές να κινηθούν ώστε να μειώσουν το κόστος, την τιμή δηλαδή, να μειώσουν την τιμή δηλαδή για να αποφελθούν από τη διαφορά. Αυτό που εννοώ είναι ότι σε αυτές, υπό αυτές τις συνθήκες κόστους υπάρχει ένα πρόσθετο πρόβλημα το οποίο προκύπτει στις ε, αγροτικές αγορές, διότι οι αλυσίδες υπερκαταστημάτων έχουν πλέον κίνητρο να μειώσουν τις τιμές ώστε να αυξήσουν τα κέρδη τους. Αυτό είναι γνωστό στην οικονομική θεωρία και ίσως όντως να ισχύει σε ορισμένους τομείς και στον αγροτικό τομέα δηλαδή. Θα προχωρήσω σε άλλη διαφάνεια. Ανέφερα πριν τις δύο δυνατότητες. Τώρα στην αριστερή πλευρά του πίνακα βλέπετε την περίπτωση, την υπόθεση δηλαδή, όπου όλες οι φίρμες αυτές έχουν το ίδιο κόστος μονάδας. 17 πένες ανά μονάδα. Επομένως η τιμή ισορροπίας στην περίπτωση αυτή είναι ότι πρέπει να είναι 17 πένες. Διότι οι γεωργοί δεν θα δώσουν χαμηλότερο κόστος και οι αγοραστές, είτε είναι ένας είτε είναι εκατό, δεν θα πληρώσουν παραπάνω. Άρα το πρόβλημα δεν προκύπτει όταν κάθε αγρότης παραγωγός έχει την ίδια μονάδα ελάχιστου κόστους, αλλά στη δεξιά πλευρά είναι η άλλη υπόθεση, η άλλη περίπτωση, όπου ορισμένες ε, ε, εταιρείες παραγωγής, ορισμένη παραγωγή δηλαδή, έχουν χαμηλότερο ε, κόστος μονάδας, 13 πένες ας πούμε, άλλο υπάρχει με 50 πένες και οι περιθωριακοί έχουν 17 πένες. Ποια είναι στην περίπτωση αυτή η τιμή ισορροπίας? Θα είναι λιγότερο από 17 πένες εφόσον υπάρχει αγοραστική δύναμη από πλευράς ε, των αγοραστών. Αυτό δείχνει η οικονομική θεωρία, διότι στην περίπτωση αυτή, αυτή της αγοράς υπάρχει κίνητρο για τους αγοραστές να περικόψουν τις τιμές κάτω από τις 17 πένες άρα ορισμένοι αγρότες θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την αγορά άλλοι θα λάβουν βέβαια λιγότερο χαμηλότερο, χαμηλότερη τιμή για τα προϊόντα τους αυτά όπως είπα λέει η θεωρία ο λόγος για τον οποίο μπορεί να υπάρχει επιπρόσθετα πρόβλημα αγοραστικής δύναμης στις αγροτικές αγορές. Κάτι που δεν ανέφερα ε, σχετικά με τη διαφάνεια είναι ότι μπορεί να καταδειχθεί και αρκετά εύκολα ότι όσο μικρότερο είναι ο αριθμός των αγοραστών, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι περικοπές των τιμών. Λιγότεροι αγοραστές θα περικόψουν την τιμή ακόμα χαμηλότερα κάτω από τις 17 πένες. Ένα από τα ερωτήματα που τίθεται βέβαια είναι ποιες δράσεις πολιτικής μπορούν να αναλυφθούν. Ας το δούμε αυτό για λίγα λεπτά. Καμία πώληση άξιων στην πραγματικότητα δεν είναι ιδιαίτερα επιθυμητή. Γιατί κανονικά θα, θέλαμε, θα προτιμούσαμε να αφήσουμε την αγορά να ρυθμίζει τα θέματα αυτά. Αν όμω υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο προκύπτει, κάποια πολιτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εδώ αναφέρω τρει στην διαφάνεια αυτή. Μπορεί κανείς να επιτρέψει στις αλυσίδες ε, ε, των σούπερ μάρκετ να συμφωνήσουν να ορίσουν υψηλότερες τιμές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, ορισμένες, ορισμένα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να αυξήσουν την τιμή του γάλακτος κατά τρία κατά τρεις πένες. Αυτό το κάνανε κυρίως για, ε, για θέμα δημόσιων σχέσεων. Το πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι μπορεί να ε, παραβιάζει την πολιτική ανταγωνισμού. Ορισμένες από τις επιχειρήσεις αυτές ε, ανακάστηκαν να πληρώσουν πρόστιμα επειδή προέβησαν σε ρύθμιση τιμών. Το άλλη, η άλλη δυνατότητα είναι να επιτραπεί στους ε, αγρότες να φτιάξουν ομάδες πολιτών Ακόμα και αν υπάρξουν όμως τέτοιες ομάδες, αυτές θα ρυθμίζουν το, την τιμή του προϊόντος τους, άρα θα λειτουργούν αυτές οι ομάδες πλέον μονοπωλιακά. Ίσως αυτό να αποτελέσει ένα αντίβαρο βέβαια στην αγοραστική δύναμη των ε, σούπερ μάρκετ, αλλά πάλι δεν είναι ιδανική λύση αυτή. Μια τρίτη λύση που περιλαμβάνω εδώ είναι η κανονιστική ρύθμιση, η ρύθμιση με, με νομοθετικό τρόπο δηλαδή, Ίσως είναι και το απλούστερο αυτό. Υπάρχουν και επιχειρήματα βέβαια κατά. Ίσως όμως είναι μια λύση εφόσον υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχουν αυτές οι τάσεις. Α, από τις τρεις αυτές βέβαια εγώ προτιμώ την τελευταία από τις αυτές λύσεις, την κανονιστική ρυθμίση δηλαδή, αλλά ίσως άλλοι έχουν άλλες απόψεις. Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε τον Ξαβιέ Ντουριέ τώρα, Γενικό Γραμματέα της Eurocommerce. Και ο τίτλος της παρουσίασης του είναι πώς μπορούν να συμβάλλουν οι έμποροι στην πιο εύρυθμη λειτουργία της ε, τροφιμικής αλυσίδας στην Ευρώπη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν να, να σας πω ότι σας ευχαριστώ για το εγχείρημα που αναλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έρχεσαι Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασφαλίσει καλύτερη λειτουργία τη αλυσίδα ευρωδιασμού στην Ευρώπη προ όφελο όλων. Θα ήθελα επίση να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το ότι έχει προσκληθεί εδώ ο τομέα του λιανικού εμπορίου στη συζήτηση. Το Eurocommerce ε, εκπροσωπεί το λιανικό εμπόριο στην Ευρώπη από τις μεγαλύτερες, τις μικρότερες ε, επιχειρήσεις ε, και ίσως καλό να ξέρετε ότι 6 εκατομμύρια εταιρείες είναι ενεργοί στο εμπόριο και το 95% είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι λοιπόν έχουμε κάποια εμπειρία σε σχέση με το εμπόριο. Επίσης 31 εκατομμύρια τομά ενεργοποιούνται στο εμπόριο και χαίρομαι που αυξάνεται ο αριθμός αυτός όμως ε, χρειαζόμαστε κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες στην αγορά προκειμένου να μπορέσουμε να αυξήσουμε τον αριθμό αυτό. Τώρα, το ιδιαίτερο στοιχείο για το εμπόριο είναι ότι έχουμε να κάνουμε με καταναλωτές ε, ε, περίπου ένα δισεκατομμύριο άτομα καταναλωτές αποφασίζουν που θα καταναλώσουν εδώ. Μιλάμε για ανταγωνισμό και θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Επίσης πρέπει να υπογραμμίσω ότι το εμπόριο ε, δεν ε, ε, ε, μάλλον έρχεται και σε επαφή με τους ε, αγρότες. Είναι αναγκαιότητα να έχουν δίκαιο εισόδημα αγρότες. Εμείς υποστηρίζουμε πλήρως, το είπε ο κύριος Μποβέ, ότι πρέπει να υπάρχει δίκαιο εισόδημα για τους αγρότες και το αξίζουν και μπορώ να σας πω ότι πρέπει να έχουμε κι εμείς ε, ένα σταθερό εισόδημα τους αγρότες για να μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό, γιατί και οι αγρότες βασίζονται σε ένα σταθερό εμπόριο. Μόνο ένας καινοτόμος τομέας μπορεί να παράσχει την γάμα φρέσκο προϊόντων που πρέπει να παράξουν οι αγρότες και που χρειάζεται και όλο εμπόριο να διανύμει ε, για να στηρίξει τη, τη ζήτηση των καταναλωτών πρέπει να δούμε ε, πώς λειτουργούν όλοι οι παράγοντες στη διατροφική λυσίδα, όχι μόνο ε, οι ε, λιανέμποροι και οι αγρότες και υποστηρίζουμε τα όσα υπόθηκαν για την εξουσία των πελετών. Δηλαδή αναφερθήκατε στο ότι ένας μόνο ε, έμπορος μπορεί να κερδίσει 10 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα. Θα ήθελα να έρθω τώρα στο θέμα των αθεμήτων πρακτικών. Στο τομέα, ο κύριος ε, Μποβέ στο έγγραφό του αναφέρεται στις καταχρηστικές πρακτικές που χρησιμοποιούν ε, οι λιανέμποροι. Λυπούμαστε για τη δήλωση αυτή, καθώς οι λιανέμποροι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν αγοράζουν από παραγωγούς δεν αγοράζουν από τους αγρότες. Εμείς ε, ε, θέλουμε, αν χρειαστεί, να αναθεωρήσουμε τη θέση μεταξύ των αγροτών και όσων αγοράζουν από τους αγρότες. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να διαφοροποιήσουμε μεταξύ των ε, καταχρήσεων της αγοραστικής δύναμης και της άσκησης της αγοραστικής δύναμης που αποτελεί τη βάση της οικονομίας της αγοράς σε οποιαδήποτε τομέα. Δεν χρειάζεται να πω, Πρόεδρε, ότι η Eurocommerce ε, είναι αντίθετη ε, στο να γίνεται κατάχρηση της αγοραστικής δύναμης, γιατί η αγοραστική δύναμη πιστεύουμε ότι ασκείται από όλους, ακόμη και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα μέρη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν αγοράζουν. Έτσι λοιπόν, υπό την σκοπιά αυτή θεωρούμε ότι οι αρμόδιες αρχέ ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν καλά τη δουλειά τους και πιστεύουμε ότι οι κανόνες περί ανταγωνισμού που υπάρχουν ε, σε εθνικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο αρκούν για να αντιμετωπίσουν τις δυσλειτουργίε τη αγορά. Ε, και μπορούμε να σκεφτούμε και περιπτώσεις όπου έχουν επιβληθεί κυρώσεις ε, και όλα αυτά μα δείχνουν ότι το σύστημα λειτουργεί. Η άσκηση της Τη ε, της αγοραστικής εξουσίας από τους λιανεμπόρους μπορεί να ωφελήσει τον καταναλωτή για τη μείωση των τιμών και όπως ε, ε, αναφέρθηκε το, το Βασίλειο έχει πει ότι γενικά η άσκηση της ε, αγοραστικής δύναμης από τους χονδρέμπορους είναι πιθανό να έχει κάποια αποτελέσματα θετικά για τον καταναλωτή, όμως ε, ε, τελικά μέσω της άσκησης της δύναμης αυτής ε, από ε, τους χονδρέμπορους. Ε, κάτι τέτοιο μπορεί να λειτουργήσει ρυθμιστικά έναντι των προμηθευτών. Σε ό,τι αφορά ε, τα προϊόντα που πρέπει να έχουμε στα ράφια ή για να από, ανεξάρτητα με το μέγεθο τους, έχουν μικρή αγοραστική δύναμη έναντι των κατασκευαστό. και εμεί θεωρούμε ότι η αγοραστική δύναμη ακόμα και των πιο μεγάλων λιανεμπόρων ε, μπορεί να υπερσκελιστεί από ε, κάποια αγαθά που ε, φέρουν μεγάλο εμπορικό σήμα. Όμως πρέπει να δούμε ποιο ασκεί την αγοραστική δύναμη και πώ μπορεί να την καταχραστεί. Και εμείς θεωρούμε ότι οι λιανέμποροι προσφέρουν ακόμη καλύτερε τιμές στους αγοραστές αν ε, δεν, θα πρόσφεραν ακόμη καλύτερε τιμέ αν δεν επιβάλλονταν κάποιε πρακτικέ από του κατασκευαστέ. Οι λιανέμποροι ναι, έχουν εισαγάγει καινοτόμα προϊόντα στην αγορά, όπω το πιο πράσινα προϊόντα και το δίκαιο εμπόριο ε, παρουσιάζουν, φέρνουν προστιθέμενη αξία για του καταναλωτέ και βοηθούν τι τοπικέ και μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει να έχουν καλύτερη πρόσβαση ε, στην αγορά, πολύ περισσότερο από ό,τι κάνουν οι κεντρικοί προμηθευτέ. Τώρα, να αναφέρω δύο λόγια σε σχέση με το θέμα του κέρδους. Η εξέλιξη των τιμών ελληνικής εξαρτάται από την τιμή που καταβάλλεται στο προμηθευτή. Ε, είπατε την Μποβέ, γιατί δεν μειώθηκαν οι τιμές σε ορισμένες περιπτώσεις. Εμείς υποστηρίζουμε αυτό που είπατε. Το και περιθώριο κέρδους των λιανμπόνων είναι 4% και δεν μπορεί να απορροφήσει ε, την αύξηση των τιμών ή να αρνηθεί τη μείωση των τιμών από αυτούς τους αγορές και φυσικά έχουμε και το πληθωρισμό ε, στο λιανικό εμπόριο, 4% όπως σας είπα. Εδώ, αν το συγκρίνετε με το πόσο κερδίζουν ε, οι ενδιάμεσοι, θα δείτε ότι κερδίζουν 3 με 5 φορές περισσότερο. Και τελικά από το λιανικό εμπόριο ε, ωφελείται ο καταναλωτής. Επίσης, εμείς βοηθούμε να μετριαστεί ο αντίκτυπος του πληθωρισμού. Αν δούμε μια πιο μακροπρόθεσμη, ακολουθήσουμε μια μακροπρόθεσμη φλουσέγγιση, θα δούμε ότι στο Βέλγιο είχαμε τα τελευταία 15 χρόνια 2% πληθωρισμό, ενώ κατά μέσο όρο ε, ο πραγματικός πληθωρισμός είχε περιοριστεί στο 1,55%. Φοβόμαστε ότι αν υπάρχει υπερβολική διαφάνεια των τιμών θα οδηγήσει σε υπερβολική γραφειοκρατία και θα εμποδίσει τον ανταγωνισμό και μάλιστα μπορούμε να οδηγηθούμε και ε, σε παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού σε σχέση με την εποπτεία που προτάθηκε από τον κύριο Μπεβέ στο ε, να παρακολουθούμε όλες τις διαδικασίες ε, των 20 ε, μεγαλύτερων πρωταγωνιστών στον τομέα. Πιστεύουμε ότι δεν είναι κάτι ρεαλιστικό, όμως υποστηρίζουμε τον κύριο Μπεβέ όταν είπε ότι η κερδοσκοπία επί των τροφίμων πρέπει να περιοριστεί. Δεν είναι προς το συμφέρον του εμπορίου να υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες. Τώρα τι μπορεί να κάνει το γύρο για να βοηθήσει τους αγρότες. Είπα νωρίτερα ότι σπανίως οι ε, ναι, αγοράζουν απευθείας από τους αγρότες. Επομένως, η δυνατότητα για ναι να βοηθήσουν τους αγρότες είναι κάπως περιορισμένες. Παρ' όλα αυτά, να σας δώσω κάποια παραδείγματα πρωτοβολιών που ελήφθησαν από τους Λιανέμπορους για να βοηθήσουν στην αύξηση του εισοδήματος γεωργών. Οι Βέλγοι ε, Λιανέμποροι πέρσι αποφάσισαν να αυξήσουν κατά 14 λεπτά ε, ε, το την τιμή του γάλακτος για τον καταναλωτή, όμως ε, το 15% του γάλακτος περνά από το λιανεμπόρο, το υπόλοιπο περνά από τη βιομηχανία. Το ότι η βιομηχανία τομέας αρνήθηκε να αυξήσει την τιμή που καταβάλλεται στον παραγωγό, ε, οδήγησε τελικά στο να υπάρχει ένας αντίκτυπος δύο λεπτών για τον παραγωγό και πολλοί ανεμπόροι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν δεσμευτεί να πληρώνουν ε, πιο πολύ από ότι η βιομηχανία. Ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο πληρώνουν 15% περισσότερο κατά μέσο όρο ε, από ότι η βιομηχανία. Και να σας πω ότι πολλοί ανεμπόροι στον τομέα των τροφίμων, προωθούν τα τοπικά προϊόντα και τον υγιεινό τρόπο ζωής και μια ισορροπημένη δίαιτα όπως και την τακτική κατανάλωση ε, των λαχανικών, φρούτων, κρέατος κτλ. Πώς μπορούμε τώρα να βελτιώσουμε τον ε, ε, γεωργικό τομέα. Πιστεύουμε ότι ο γεωργικός τομέας σε πολλές χώρες στην Ευρώπη χαρακτηρίζεται ακόμη από κατακαιρματισμό και αναποτελεσματικότητα. Το να δημιουργηθούν οργανώσεις παραγωγών σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση των αγροτών έναντι των μεταπητών και αναρωτιόμαστε αν ο κανονισμό 1234 1234-2007 πώς θα μπορούσε να επεκταθεί ε, να καλύπτει και τα προϊόντα ε, τα γαλακτοκομικά πέρα από το λάδι, παραδείγματο χάρη. Ε, τώρα έχουμε μία επιτυχία που σημειώθηκε στα βιολογικά τρόφιμα και στο μεγαλύτερο μερίδιο που αρχίζουν να καταλαμβάνουν στην αγορά. Αυτό μας δείχνει ότι οι καταναλωτές για να έχουν καλύτερη ποιότητα στα τρόφιμα πληρώνουν περισσότερο. Επίσης, σε πρόθεση ε, των τοπικών ε, προϊόντων, ε, κάτι τέτοιο, θα μπορούσε να ενδυναμώσει τη θέση των αγρότων στην αγορά και έχουμε και την κάθετη ένταξη. Το αναφέρετε και εσείς αυτό, γιατί παίρνουν το σχάρι δεν θα μπορούσαν να πουλούν η παραγωγή απευθείας στον καταναλωτή. Αν φυσικά γνωρίζουμε ότι πληρούνται και τα ίδια κριτήρια ποιότητας ευσήμανσης συχνηλασιμότητας. Οποιοδήποτε μέτρο που μπορεί να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθήσει του αγρότε να σταθεροποιήσουν ε, το εισόδημό του. θα ήταν ευπρόσδεκτο συμπερασματικά. Πιστεύουμε ότι αξίζουν ένα δίκαιο εισόδημα και σταθερό εισόδημα οι οργοί. Θα πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση των αγροτών στη χρηματοδότηση. Αυτό που προτείνουν ο κύριος Δεσούτερ και ο κύριο Μποβέ, δηλαδή μείωση τη κερδοσκοπία θα πρέπει να εξεταστεί και φυσικά οποιαδήποτε κατάχρηση ε, στον τομέα τη αγοραστική δύναμη. θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Φυσικά εδώ διαφαίνεται η αναγκαιότητα τα να δούμε πού προέρχονται οι καταχρήσεις αυτές. Η ανάγκη της διαφάνειας ε, θα πρέπει να τηρείται καθ' όλη την αλυσίδα, όμως η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνει χωρίς να υπάρχει προς το διοικητικό άχθος και φυσικά πάντοτε θα πρέπει να τηρείται και το επαγγελματικό απόρριτο. Οι αρχές ανταγωνισμού πρέπει να διασφαλίσουν ε, ότι αυτό το εγχείρημα δεν οδηγεί σε καταχρήσεις και να κλείσω εδώ οι αθέμητες πρακτικές ή πρακτικές που στρέφονται κατά την αρχή, της αρχής της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να διευρυνθούν και να επιβληθούν κυρώσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και με αυτή την παρουσίαση κλείσαμε τον πρώτο γύρο των τοποθετήσεων. Ο κύριος Αλμπερντές. Ευχαριστώ. Χαίρομαι για την διεξαγωγή της παρούσας ακρόασης. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον συνάδελφο Μποβέ. Έγραψε μια έκθεση που με βρίσκει σε μεγάλο βαθμό σύμφωνο. Θα κάνουμε ορισμένες τροποποίησεις σε κάποιες διατυπώσεις και σε ορισμένα περιορισμένα θέματα ουσίας, αλλά ομολογώ ανοιχτά και καθαρά ότι δεν θα συνέτασα πολύ διαφορετικά την έκθεση αυτή. Τώρα, έρχομαι σε ορισμένα από όσα συζητήθηκαν προηγουμένως. Ένα θέμα θέλω να θίξω πρώτα, κύριε Μποβέ. Θα πρέπει να ζητήσουμε στην έκθεση η προθεσμία πληρωμής για τα τρόφιμα να είναι της τάξης των 30 ημερών. Αυτό θα ε, βοηθήσει και θα συμβάλλει δηλαδή και στη βελτίωση της κατάστασης των αγροτών. Τώρα, αυτά για τα discount και τα λοιπά, εγώ ως αγρότης δεν έχω έρθει εδώ για να υπερασπιστώ αυτά τα πράγματα, αλλά και έχω υπόψη μου τη γερμανική κατάσταση, δεν γνωρίζω η κατάσταση πως είναι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά ψήφισαν στην ουσία οι καταναλωτές με τον τρόπο που πηγαίνουν και ψωνίζουν. Η πεθρά μου είχε ένα μικρό κατάστημα σε ένα χωριό και αναγκάστηκε να το κλείσει γιατί ο κόσμος δεν πήγαινε πλέον να ψωνίσει εκεί, πήγαιναν στο σούπερ μάρκετ και στα λιγόμενα discount stores που προσφέρουν μεγάλες εκπτώσεις και που το 95, το 1995 δηλαδή ήταν στο 27% και σήμερα έχουν φτάσει στο 55% του συνόλου ε, του όγκου κατανάλωσης απεφάσισαν εν τέλει δηλαδή οι καταναλωτές που θα πάνε να ψωνίσουν. Και αυτό δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Ένα ωστόσο μπορούμε να διαπιστώσουμε. Ίσως είναι διαφορετικά τα πράγματα σε άλλες χώρες. Πάντως στη Γερμανία οι μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων μετακύλησαν το όφελος από την μείωση των τιμών στους καταναλωτές. 20% μείωση τιμών που πάει στον καταναλωτή. Εποφελεί το καταναλωτής δηλαδή. Σε μεγάλο βαθμό, 20% μέχρι και 35% έχουν ωφεληθεί από τέτοιες περικοπές τιμών οι καταναλωτές. Και οι καταναλωτές δαπανούν όλο και λιγότερο ποσοστό του εισοδήματό του για την αγορά τροφίμων. Έχουμε φτάσει στο σήμερα στο 12% του εισοδήματό του να πηγαίνει στην αγορά τροφίμων, ενώ το 60% ήταν 40%. Ένα πράγμα λοιπόν θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο. Και ε, στην αγορά τροφίμων υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Εγώ είμαι και πρόεδρος ενός μεγάλου συνεταιρισμού γαλακτοπαραγωγών. Για τα μέλη μας αυτά θέλουμε βεβαίως τις βέλτιστες συνθήκες διάθεσης του προϊόντος στην αγορά. Το κέρδος μας είναι μοναχά 0,2% στην, ε, στον συνεταιρισμό μας αυτό. Όλα τα υπόλοιπα πηγαίνουν στους παραγωγούς, στον παραγωγό. Κάθε κέρδος πηγαίνει στον παραγωγό. Δεν μπορούμε όμως να προσφέρουμε και φθηνότερα. Ούτε μπορώ να μεμφθώ το εμπόριο, διότι και το εμπόριο συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο. Εάν μια μεγάλη φίρμα χρειάζεται για παράδειγμα 10.000 λίτρα καυσίμου, πηγαίνω σε άλλο, σε άλλο είδος προϊόντος, θα ζητήσει 10 προσφορές από, τους, ε, από αυτούς που προσφέρουν στην αγορά ε, καύσιμα και θα επιλέξει τη φθηνότερη. Το ίδιο γίνεται και για το τρόφιμο. Κάτι που με ενοχλεί βέβαια περισσότερο και εκεί φαίνεται βέβαια καθαρά η αγοραστική δύναμη κάποιων ομήλων όταν γίνονται για παράδειγμα προσπάθεια μείωσης του κόστους της συσκευασίας. Αλλάζει η συσκευασία του ε, γάλακτος για παράδειγμα για να γίνει πιο φθηνό εν τέλει για τον τελικό καταναλωτή. Το κάναμε εμεί αυτό, αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε τι συσκευασίε και μα κόστησε συνολικά στο συνεταιρισμό μα δηλαδή 700.000 ε, ευρώ. Έρχονται καμιά φορά τα σούπερ μάρκετ και λένε έχετε δύο μήνες προθεσμία για να αλλάξετε τις συσκευασίε. Αυτό όντως είναι ε, μια επίδειξη της αγοραστικής τους δύναμης. Στην Ευρώπη βέβαια είναι διαφορετικές οι καταστάσεις. Για παράδειγμα η τιμή του γάλακτος. Δεν γνωρίζω ποια είναι η σωστή τιμή του γάλακτος. Δίπλα μου εδώ κάθεται ο συνάδελφός μου κύριος Ντόρφμαν. Εμείς στέλνουμε γάλα από τη Βαβαρία στην Ιταλία. Στο νότιο Τυρόλο η τιμή του γάλακτος του λίτρου είναι 50, 50 λεπτά. Παρόλο που από τη Γερμανία φεύγει με τιμή 32 λεπτά. Εν τέλει όμως αποφασίζει ο κόσμος, ο πληθυσμός του Νότιου Τυρούλου. Αποφασίζουν ότι θέλουν να αγοράσουν γάλα του Νότιου Τυρούλου. Και επομένως το πληρώνουν, είναι να το πληρώσουν και περισσότερο. Ενώ από τη Γερμανία και την Αυστρία θα μπορούσαν να ε, αγοράσουν φθηνότερο γάλα. Δεν αλλάξουμε και τίποτα εκεί. Τα αυτοκίνητά μας λοιπόν περνάνε μέσα από τον Νότιο Τυρόλο χωρίς να ξεφορτώσουν και συνεχίζουν προς Ιταλία με τα 32 λεπτά. Και βλέποντας τι γίνεται και στη Βόρεια Γερμανία, πάνω στην Βόρεια Θάλασσα, εκεί είναι διαφορετικές οι τιμέ Α έχουμε σαφώ υπόψη ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει μια απόλυτα δίκαιη τιμή για όλου. Και ακόμα ένα σύντομο σχόλιο. Θεωρώ ότι η αγορά θα ρυθμίσει ορισμένα πράγματα. Στο περιβάλλον μου διαπιστώνω ότι ένα μέρος των γεών δεν χρησιμοποιείται πλέον για την παραγωγή ε, γεωργικών προϊόντων, δηλαδή για την παραγωγή τροφίμων. Αρχίζουν ορισμένα εδάφη και ε, χρησιμοποιούνται για την παραγωγή καυσίμων αν συνεχίσουν τα πράγματα έτσι, θα, συνεχίσει, θα, θα αρχίσει έτσι να κινείται ο παραγωγός. Και αν κάποια στιγμή αυξηθούν οι τιμές των καυσίμων, τότε ο Γιώργος θα ε, κερδίζει περισσότερα ε, παράγοντας ε, φυτά για καύσιμα από ότι ε, με τα τρόφιμα και επομένως θα απαλλαγεί και από οποιασδήποτε εξαρτήσεις που έχει από επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι η αγορά θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Αυτό που με ενοχλεί είναι η κατάσταση όπως διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή, διότι υπάρχουν αγρότες οι οποίοι βρίσκονται σε δινή θέση. Πρέπει να αλλάξουν ορισμένα πράγματα ώστε να παραμείνει η γεωργική παραγωγή εκεί που γίνεται και διεξάγεται αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι τον κύριο Μποβέ για την έκθεσή του. Ο κύριος Καπουλασάντος στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ε, παρουσιάσεις σας. Όμως νομίζω ότι εδώ εμείς πρέπει να επικεντρωθούμε στο ουσιαστικό ζήτημα. Εγώ άκουσα τον εκπρόσωπο της Eurocommerce ο οποίος εκπροσώπησε τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, μας τους παρουσίασε σαν θύματα αυτής της διαδικασίας. Όμως, εγώ νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στο κεντρικό ζήτημα. Δηλαδή, το το δικό μας κοινωνικό μοντέλο έχει θέσει σε μια πολύ δύσκολη θέση τους παραγωγούς έναντι των μεγάλων σούπερ μάρκετ και το πρόβλημα που μας τίθεται είναι ότι εδώ έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία προωθεί την ελεύθερη αγορά, το ελεύθερο εμπόριο. Πώς ε, μπορούμε να παρέμβουμε υπέρ του αδύναμου κρίκου της αλυσίδας γιατί τελικά ε, βλέπουμε ότι εδώ η αγορά από μόνη τη δεν επιλύει το πρόβλημα, αλλά αυτό επιδεινώνει και εμείς ε, εδώ ίσως πρέπει να αλλάξουμε το βασικό κανόνα λειτουργίας της κοινωνίας μας. Η δική μας είναι ότι αν δεν έχουμε κάποια παρέμβαση στην αγορά τελικά το πρόβλημα δεν μπορεί να επιληθεί υπέρ των γεωργών και εμείς τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή τη συζήτηση, να προσπαθήσουμε να δούμε πώς είναι δυνατόν να παρέμβουμε στην αγορά χωρίς ε, να ε, δημιουργήσουμε πρόσκομα στον ελεύθερο ανταγωνισμό και εγώ δεν νομίζω ότι δίνεται απάντηση μέσω της έκθεσης του κυρίου Μπαβέ, ούτε οι λύσεις που μας παρουσιάστηκαν μέχρι τώρα είναι αισιόδοξε. Άκουσα τον κύριο Τσούτερ, ο οποίος παρουσίασε ως λύση την τοπική γεωργία και τις τοπικές αγορές, όμως όλοι γνωρίζουμε ότι η παραγωγή είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και χρησιμοποιούνται μηχανήματα κυρίως στην παραγωγή ε, και δίχως τέτοιου είδους παραγωγή η κοινωνία μας δεν θα μπορούσε να επιβιώσει. Έτσι λοιπόν το συμπέρασμα που εξάγω είναι ότι για το πρόβλημα αυτό δεν μπορούμε να βρούμε τομέακες λύσεις. Ε, εγώ νομίζω ότι η λύση πρέπει να είναι πολιτική, δεν μπορεί η αγορά να επιλύσει το θέμα και οι πολιτικοί πρέπει να συνεισφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή δεν έχω το μαγικό ραβδί για να επιλύσω το πρόβλημα, αλλά έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι αν δεν υπάρχει παρέμβαση στους κανόνες της αγοράς, ε, τίποτα δεν μπορεί να γίνει και η απόφαση αυτή μπορεί να ληφθεί μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαφορετικά δεν θα υπάρξει λύση του προβλήματος γιατί η λύση στην οποία βρίσκονται η παραγωγή αφενός και οι οποίοι ε, μαζικά αποκτούν και διανέμουν τα προϊόντα τους από την άλλη. Είναι μια κατάσταση ανισορροπίας ε, και εγώ δεν νομίζω ότι η αγορά μπορεί να επιλύσει το θέμα αυτό, ούτε μέσω της των κινήτρων που δίνονται για την ε, προσφορά. Έτσι λοιπόν πρέπει να βρούμε μια λύση που να περνά από την ε, παρέμβαση στην αγορά χωρίς φυσικά να διακυβεύουμε την ελεύθερη διακίνηση των αγαθών ούτε το οικονομικό μας σύστημα στο οποίο έγκυται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι μπορούν να θέσουν και ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες, αν το επιθυμούν. Κύριε Λάλη. Uh, Λίγα σχόλια σχετικά με τις παρεμβάσεις που ακούσαμε προηγουμένως. Βρήκα ενδιαφέρουσες τις απόψεις του Ρότζερ Κλάρκ σχετικά με την πρόταση για, την, για τον διορισμό ενός ombudsman και ένα θέμα που θα μπορούσε να εξεταστεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί οι μεγάλες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου είναι όντως συχνά πολυεθνικές. Σχεδιάζεται τέτοιος θεσμός στο Ενωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία. Για μένα πάντως μου φαίνεται ουσιώδες να εξεταστεί η λύση αυτή. Χρειάζεται και ένας κώδικας που να είναι νομικά εξαναγκαστός, δηλαδή να μπορεί να επιβληθεί. Θα με ενδιαφέρει επίσης να ακούσω τις απόψεις σχετικά με διαφάνεια και με το λεγόμενο naming and shaming, δηλαδή να ανακοινώνονται τα ονόματα των παραβατών ή των παραβατριών εταιριών. είναι και γεγονό ότι ε, διαμορφώνονται σε υψηλότερα επίπεδα τα κέρδη του όταν αυξάνονται οι τιμές. Εποφελούνται επομένω. Άρα είναι ε, χρήσιμο να γίνονται γνωστοί. Κύριος Ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις και στον κύριο Ντεσούτερ που εξήγησε ότι ο ρόλος της γεωργίας είναι σημαντικός και παγκόσμια και η αδυναμία της είναι και παγκόσμια. Είναι γεγονός ότι ο πιο αδύνατος κρίκος της αλυσίδας στην προμήθεια τροφίμων είναι η αγροτική παραγωγή. Υπάρχουν βέβαια διαφορετικές δομές. Το πρώτο θέμα το ξεκαθάρισε ο Ζωζέ Μποβέ στην εκθεσή του. <clears throat> Ότι δηλαδή χρειαζόμαστε διαφάνεια στην αγορά, την οποία δεν έχουμε ακόμα. Δεν γνωρίζουμε και τι είναι απαραίτητο να γίνει, διότι όπως είπα δεν υπάρχει διαφάνεια. Άρα πρέπει να βγουν τα πράγματα καθαρά στη δημοσιότητα. πρέπει να γίνουν διαφανείς και οι πρακτικές. Δεν μπορούμε να μιλούμε για διαφανή ανταγωνισμό όταν σε πολλές χώρες ρυθμίζουν στην ουσία την αγορά του αγροτικού προϊόντος ορισμένοι όμιλοι. Ε, πάρουμε αρκετά σοβαρά το θέμα, μιλούμε για παράδειγμα πολύ για τις άμεσες ενισχύσεις οδήματος των παραγωγών. Το ζήτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε και στο εμπόριο που θα είναι πολύ καλύτερο παρά να δίνουμε άμεση ενίσχυση 30, 300 400 ευρώ ανά εκτάριο στον παραγωγό. Για τον δεύτερο παρεμβαίνοντα ήθελα να ρωτήσω εάν αρκεί μια οικειοθελής λύση του είδους ombudsman ή κώδικα διοντολογίας αρκούν τέτοιες λύσεις. Δεν νομίζει ότι χρειάζεται να προχωρήσουμε περισσότερο και να επιβάλλουμε νομοθετικά λύσεις. Άλλη ερώτηση. Ο εκπρόσωπος του λιανικού εμπορίου είπε ότι έχει γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια προώθησης ε, δίκαιου εμπορίου και δίκαιων προϊόντων. Μα είναι είναι σωστό να γίνει μια ρύθμιση εκ των άνω και όχι από το ίδιο το εμπόριο. Πρέπει να αναζητηθούν δυνατότητες να επιβληθούν νομοθετικές ρυθμίσεις και όχι να περιμένουμε από το ίδιο το εμπόριο να αυτορυθμιστεί. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε νομοθετική ρύθμιση για να προχωρήσει και το έντιμο, το δίκαιο εμπόριο, το fair trade. Και κάτι ακόμα για τις δημόσιες προμήθειες εφόσον υπάρχει δημόσια αγοραστική δύναμη και σημαντική μάλιστα, πρέπει αυτή να έχει υποδειγματικό ρόλο, ρόλο προτύπου. Και ιδίω για τους οργανισμούς εκείνους οι οποίοι προσφέρουν και διατροφή να τηρούν αυστηρά τις ε, διατάξεις περί δημοσίων προμηθειών, ε, περί διαγωνισμών κλπ. Και όχι και βεβαίω να βάζουν και άλλα κριτήρια και όχι μόναχα το πιο συνοφθηνότερος. Εν τέλει, θα πρέπει να προκύψουν συμπεράσματα από τη συζήτηση αυτή, τα οποία να ενισχύσουν την θέση του παραγωγού μέσα στην αλυσίδα προμήθειας τροφίμου. Και να μην αρκεστούμε μονάχα σε συστάσεις. Πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα συμπεράσματα. Vă mulțumesc. Are cuvântul în continuare domnul Alve. Ο κύριος Αλντές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ συζητάμε ένα θεμελιώδες ζήτημα γιατί προσανατολίζουμε την αγροτική πολιτική προς την αγορά και προσανατολίσουμε προς ε, την αγορά και με αυτόν τον τρόπο η αξία που έχει αγορά είναι όλα ένα και πιο καθοριστική για τους παραγωγούς. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς συμπεριφέρονται οι αγορές σήμερα. Οι τιμή στις αγορές καθορίζονται από τους καταναλωτές. Ο καταναλωτής λέει πόσο θέλει να πληρώσει για τα συγκεκριμένα προϊόντα και ο διανομέας είναι αυτός που λαμβάνει αυτό το ποσό και καταρχήν είναι αυτός ο οποίος ε, θα διανέμει στην υπόλοιπη αλυσίδα το ποσό αυτό. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε εδώ πώς συμμετέχει ο διανομέας και ποιο θα είναι το εισόδημα που θα δοθεί τελικά στο παραγωγό. Και φυσικά ε, όλα αυτά πρέπει να τα αναλύσουμε. Και γι' αυτό πρέπει να παρατηρήσουμε τα στοιχεία αυτά με πάσα διαφάνεια και γι' αυτό πρέπει να επαληθεύσουμε, να δούμε ποιες είναι οι πρακτικές που υπάρχουν σε αυτό το συσχετισμό, ποιες είναι οι ανταγωνιστικές πρακτικές και σε ποιο βαθμό σέβονται το ε, δίκαιο του ανταγωνισμού που υπάρχουν σήμερα, γιατί πάρα πολλά προβλήματα που αναφέρθηκαν εδώ θα μπορούσαν να λυθούν μέσω της νομοθεσίας. Εμείς πολλές φορές ε, δεν έχουμε την ε, ικανότητα να εποπτεύσουμε, ε, παίρνοντα χάρη, μία, ένα τομέα διανομής, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εξουσία και σήμερα, ούτε καν τα εθνικά εργαλεία δεν μπορούν να αξιολογήσουν ορθά τις πρακτικές αυτές. Γι' αυτό θα έπρεπε να δημιουργήσουμε ένα κοινοτικό οργανισμό, γιατί μιλάμε για πρακτικές που πρέπει να ρυθμίζονται σε επίπεδο ένωσης, γιατί είναι παγκόσμια η αγορά και μιλάμε και για εσωτερική εσωτερική αγορά δεν πρέπει να έχουμε κατακαιρματισμό ε, σε κώδικες ε, βελτίστων πρακτικών σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν η παρακολούθηση αυτή να γίνεται σε όλα τα επίπεδα και θα πρέπει να δούμε τι πρακτικές εφαρμόζονται για ορισμένα προϊόντα. Θα πρέπει να δούμε τι τιμή πληρώνεται στον παραγωγό και μάλιστα αυτό για πολύ σημαντικά προϊόντα όπως είναι το γάλα, όπως είναι το ρύζι. Και ε, νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε. Επίσης, πώς μπορούμε σήμερα να επιτρέπουμε ένας διανομέας να έχει και δικό του σήμα και να μπορέσει να ρυθμίσει το που τοποθετούνται τα σήματα αυτά, δηλαδή και να μπορεί να καθορίσει πού θα μπει στο ράφι το προϊόν, πώς θα είναι η συσκευασία, τι ε, προσφορές θα κάνει. Νομίζω ότι αυτό ούτως ή άλλως έχει επίπτωση στο εισόδημα ε, των υπολείπων στην αλυσίδα και κυρίως στο εισόδημα του παραγωγού. Έτσι λοιπόν αυτά θα πρέπει να τα δούμε στα πλαίσια της ρύθμισης που εξετάζουμε. Σας ευχαριστώ. Thank you, Chairman. Κυρία Μαγκίνες, να ξέρω ότι περνά ο χρόνος. Έτσι λοιπόν ε, θα ήθελα να κάνω κάποιες σκέψεις και θα ήθελα να τις σχολιάσετε γιατί εμπλέκομαι στην ομάδα που συζητά ακριβώ αυτό το θέμα. Τι πιστεύετε για τις ιδέες που προέρχονται από τους παραγωγούς και έχουν να κάνουν με τα σούπερ μάρκετ. Καταρχήν, ότι πρέπει να υπάρχει ένα όριο σε σχέση με το μερίδιο αγοράς ε, για κάθε συγκεκριμένο όμιλο γενικό εμπόριο 20% δηλαδή ε, του μεριδίου της αγοράς και για να εξηγήσω, λένε η παραγωγή, ότι αν δεν είχαμε τόσο μεγάλη συγκέντρωση με τόσους λίγους παίκτες, ε, τότε θα μπορούσαν περισσότεροι να πουλήσουν τα προϊόντα τους και αυτό θα ήταν καλύτερο για τους καταναλωτές, παρά το αντίστροφο. Δεύτερον, ε, ακούστηκαν ε, κάποιοι να τοποθετούνται για αυτές τις ιδιωτικές σημάνσεις. Εγώ πιστεύω ότι ε, εξακολουθεί να υπάρχει προσθεμένη αξία για τους παραγωγούς. Όμως τι σκέφτεστε αν απαγορεύουμε αυτές τις ιδιωτικές σημάνσεις στον διατροφικό τομέα. Μπορείτε να απαντήσετε σε αυτά τα συγκεκριμένα σημεία παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δανέλης. Κύριε Πρόεδρε, όλοι συμφωνούμε ότι ο παραγωγός εκτίθεται στην αγορά και καλείται να κερδίσει το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματό του, αν όχι ολόκληρο, από την αγορά. Όμως τι συνθήκες επικρατούν στις αγορές που καθορίζουν τελικά το εισόδημα του παραγωγού, αυτό είναι που μας απασχολεί. Πρώτο, στις αγορές γεωργικών προϊόντων παρατηρείται εξαιρετική αστάθεια που στο μέλλον μπορεί και να ενταθεί περαιτέρω εξαιτίας και της κλιματικής αλλαγής. Δεύτερο, στις αγορές εμπορευμάτων, γεωργικών ενέργειας και ορυκτών μετάλλων που επηρεάζουν το κόστος γεωργικής παραγωγής, οι τιμές έχουν εκτοξευθεί στα ύψη τα τελευταία χρόνια. Και τρίτο, στην αγροδιατροφική αλυσίδα οι επιχειρήσει λιανεμπορίου επεκτείνονται συνεχώς σε βάρος του παραγωγού, ο οποίος χάνει συνεχώς διαπραγματευτική δύναμη και πολλές φορές γίνεται και θύμα αθέμητων πρακτικών. Στις δύο τελευταίες κατηγορίες έχει αναγνωριστεί και από την ίδια την Επιτροπή τουλάχιστον έλλειμμα διαφάνειας. Να απαιτήσουμε λοιπόν σωστά από τον παραγωγό να προσαρμοστεί στις απαιτήσει αγοράς. Αλλά αυτό είναι δίκαιο μόνο αν έχουμε εξασφαλίσει ότι η αγορά λειτουργεί με διαφάνεια και σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, διότι διαφορετικά θέτουμε εσκεμένα και σε γνώση μας τον αγρότη ενώπιον μιας ισοπεδωτικής, αθέμητης κατάστασης και μάλιστα τον εγκαταλείπουμε εκεί άοπλο. Η Επιτροπή έχει ήδη χαράξει ένα οδικό χάρτη για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγροδιατροφικής αλυσίδας, αλλά το πρόβλημα είναι άμεσο και πιεστικό και οι διαδικασίες οι οποίες προτείνει η Επιτροπή είναι χρονοβόρες και ίσως και αμφιβόλου αποτελεσματικότητας. Προτείνει για παράδειγμα μεταξύ άλλων ενίσχυση ανταγωνιστικότητας της αγροδιατροφικής αλυσίδας μέσω της ενθάρρυνσης στη δημιουργία οργανώσεων παραγωγών Μα έχουμε αποτύχει ως Ευρωπαϊκή Ένωση τη λειτουργία αυτού του θεσμού και αυτό είναι μείζον πρόβλημα διότι οι οργανώσεις παραγωγών αποτελούν θεωρητικά τουλάχιστον τη λύση πολλών από τα προβλήματα του μικρομεσαίου παραγωγού και του ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου. Ή προτείνει χρόνο για να κατανοήσει τη λειτουργία της αλυσίδας ανακράτος μέλος. Να το κάνει. Αλλά εντωμεταξύ κάτι πρέπει να γίνει γιατί δεν μπορεί ο παραγωγός να συνεχίζει να εκτίθεται σε μη ανταγωνιστικά περιβάλλοντα και να τους δείτε να λειτουργεί ανταγωνιστικά. Είναι κρίσιμο επομένως να γίνουν δύο πράγματα. Πρώτο, να ληφθούν διαφορετικά μέτρα που να καλύπτουν όλο το χρονικό φάσμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, γιατί χρειάζονται άμεσα μέτρα ανακούφισης μέχρι να ληφθούν μακροπρόθεσμα, εκείνα δηλαδή τα μέτρα ριζικής αντιμετώπιση των προβλημάτων. Και δεύτερο, τέλος, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη λειτουργία των ομάδων παραγωγών. Πρέπει να δούμε γιατί δεν έχει επιτύχει αυτός ο θεσμός και να προβούμε το συντομότερο δυνατό σε βελτιωτικές ενέργειες για την επίλυση των προβλημάτων, αλλά συνολικά σε κοινοτικό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα σήμερα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και θέλω να σταθώ σε δύο επίπεδα, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, και να διαπιστώσω ότι αν το κέρδος είναι κάτι το υγιές στην οικονομία, η αναζήτηση του ανωτάτου κέρδους είναι το κακό πράγμα της οικονομίας και δηλητηριάζει την όλη αλυσίδα. Η πίεση που ασκείται από την διανομή και όχι μόνο από τη μεταπητική βιομηχανία, για αυτούς μιλάμε λίγο, διότι ξέρουμε ότι αναζητούν αναζητούν τη, λύση για το γάλα, αλλά θα έπρεπε και αυτοί να εκπροσωπούνται εδώ. Τώρα για τον κύριο Κλάρκ, σε ευρωπαϊκό επίπεδο λέει ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια καλύτερη ρύθμιση των αγορών. Αυτό το οποίο δολοφονεί σήμερα τη Γεωργία είναι αυτή η τρομερή αστάθεια των τιμών που όπου ο Γιωργός δεν ανταμείβεται πλέον για την εργασία του. Το 70% των γεωργών στην περιοχή μου Συγγνώμη, το, το, οι γεωργοί στην περιοχή μου με 70, παίρνουν 70% επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 30% μόνο από τη δουλειά τους. Είναι κάτι το αναξιοπρεπές αυτό. Θα πρέπει να μείβονται για τη δουλειά τους. Η, η γεωργία ε, παίζει η παραγωγή ανάλογα με τις χρονιές, το ξέρουμε. Έχουμε καλές χρονιές ε, και καλή χρονιά παραγωγής επιτρέπει ε, στον παραγωγό να επιβιώνει σε χειρότερες χρόνιες. Να έχουμε μηχανισμούς λοιπόν αποθήκευσης και ντεστοκάζ ανάλογα με τις χρονιές. Το είχαμε και στο παρελθόν αυτό όπου το σύστημα λειτουργούσε σαν ένα φίδι σε ένα τούνελ. Λοιπόν, τι λέει ο κύριος Κλάρκ, πρέπει να το ρυθμίσουμε αυτό ή όχι. Λοιπόν, είναι αυτανόητο τώρα ότι ο Ζωζέ Μποβέ έκανε καλή δουλειά, αλλά για τον κύριο Σκούτερ εγώ θέλω να μιλήσω, ο οποίος έχει κάνει πολύ σωστή εργασία στον ΟΗΕ. Ήταν πολύ σωστά αυτά που μας είπε. Οι μηχανισμοί κερδοσκοπίες ε, στους, ε, στα τρόφιμα είναι κάτι το οποίο σοκάρει. Αλλά μήπως θα έπρεπε να ανατρέψουμε την τάση. Εγώ δεν άκουσα σήμερα να γίνεται αναφορά στην ΠΟΕ να βγάλουμε από την ΠΟΕ τα γεωργικά προϊόντα, ναι ή όχι. Και η ΠΟΕ μήπως κάνει λάθος στρατηγική για να όταν θέλει να αλλάξει το σύστημα και πιστεύει ότι το παγκόσμιο εμπόριο θα αλλάξει την κατάσταση. Ξέρουμε ότι έχουμε ένα δισεκατομμύριο κόσμο ο οποίος ε, τρέφεται άσχημα, εκ των οποίων μέγα μέρος είναι γεωργοί οι ίδιοι. και Μία κοινή λήψη θέσης όλων των πρωταγωνιστών της αλυσίδας θα μπορούσε να μας βοηθήσει ε, καταρχήν ε, εγγυόμενη αυτάρκεια και αυτοκατανάλωση στις αναπτυσσόμενες χώρες πριν αρχίσουμε δηλαδή και να σταματήσουμε τέλος πάντων αυτήν την ιστορία με την ανθρωπιστική βοήθεια όπου εμείς περνάμε, ε, πηγαίνουμε τα τρόφιμα από τη μια στην άλλη άκρη του πλανήτη. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω εγώ το λόγο στον εκπρόσωπο της ΟΚΕ, τον κύριο Νάρο. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ την Επιτροπή Γεωργίας που επιτρέπει στην ΟΚΕ να μοιράζεται μαζί σας τις σκέψεις μας για ένα πρωταρχικό θέμα πώς πρέπει να γίνεται η όλη αναλογία ε, του κόστους ε, στην αλυσίδα. Εγώ λέγομαι Πέδρο Νάρο και είμαι εισηγητής ε, για το αντίστοιχο θέμα στην ΟΚΕ. Η έκθεση της ΟΚΕ είναι σε φάση επεξεργασίας. Αλλά για τον ίδιο λόγο και εμείς οργανώνουμε μια μεγάλη διεθνή διάσκεψη στη Βαλένσια φυσικά ο, στις, ε, δύο, στις 4 ε, Ιουνίου με την ενίσχυση του Κοινοβουλίου. Εμείς θέλουμε να έχουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο Ξέρουμε, θέλουμε να έχουμε καθαρούς ε, κανόνες του παιχνιδιού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεσμευτεί να, εναρμόσει, εναρμονίσει την ομοθεσία και είμαι υπέρ του να ληφθούν μέτρα και γιατί να μην το πω πολλές φορές δεσμευτικά. Οι περισσότεροι από εδώ σήμερα που παρακολουθούν αυτή τη συνάντηση συμφωνούν με τις αναλύσεις της Κομισιόν στα διάφορα έγγραφα. Δεν είναι ούτε ένα ούτε δυο, πολλά έγγραφα είναι. Για τις τιμές, για την αλυσίδα, για τα επίπεδα υψηλού επίπεδου. Και όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε στην περιγραφή της κατάστασης από την Κομισιόν. Θα πρέπει λοιπόν στη Βαλένσια πέρα από την, την εξέταση όλης της αλυσίδας θέλουμε να εξετάσουμε τους δύο αδύναμους κρίκους, τους γεωργούς και τους καταναλωτές. Πρέπει να περάσουμε στη δράση. Φτάνει με μελέτες, εκθέσεις, θέλουμε να έχουμε μέσα, θέλουμε μέτρα να εξισορροπήσουν την κατάσταση διότι έχουμε μία συζήτηση που είναι πλέον εγκάρσια για την ε, γεωργία, για την ε, αλυσίδα. Είναι μία συζήτηση πολύ πιο βαθιά, όπως έλεγε και ο κύριος Μποβέ, τι η γεωργία θέλουμε εμείς για την Ευρώπη. Πρέπει να την επιλέξουμε. Υπάρχουν τρία βασικά σημεία για μας ε, στην, στο θέμα της τροφιμικής αλυσίδας. Είναι πώς μπορούμε να έχουμε καλές ε, σχέσεις ε, ε, στην αγορά τροφίμων. Θέλουμε συμβόλαια, θέλουμε να έχουμε κώδικου και καλή συμπεριφορά, θα επιβραδεύουν τους καλούς, θα τιμωρούν τους κακούς. Θέλουμε όμπουσμαν. Ή τέλος πάντων ένα ελεγκτικό όργανο. Το δικαίωμα του ανταγωνισμού πρέπει να διαφοροποιηθεί σε εθνικό επίπεδο και να εναρμονιστεί σε ευρωπαϊκό. Θα τα πω ακόμη πιο γρήγορα γιατί έχω ελάχιστο χρόνο, λέει ο μιλτής Διαφάνεια σημαίνει παρατήρηση των τιμών. Πρέπει να έχουμε μέσα για να αντιδρούμε γρήγορα και αποτελεσματικά αλλά και ευέλικτα όταν έχουμε αυξήσει των τιμών που είχαμε τα τελευταία χρόνια στην αγορά. Τελευταίο, πώς να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα. οργανώσεις ε, παραγωγών σύμφωνοι αλλά λειτουργούν αποτελεσματικά, εξυπηρετούν τον παραγωγό, είναι αποδοτικές. Όπως είπε δηλαδή και ο Έλληνας ομιλητής, πρέπει να τα βελτιώσουμε όλα αυτά. Και τελευταίο, να επισημάνω το θέμα της απορρίθμισης των αγορών που μας οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Ο κύριος Κάπουλα Σάντος έλεγε ότι υπάρχει απεσιοδοξία και εγώ αισιόδοξο όμως είμαι Φτάνει να ληφθούν μέτρα, μέτρα τα οποία δεν είναι μόνο δημοσιονομικά μέτρα. Χρειάζεται μία πολιτική που θα ενισχύσει ουσιαστικά την τροφιμική αλυσίδα. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε το πρώτο μέρος της συζήτησης να απαντήσουν σύντομα ελπίζω οι εμπειρογνώμονες γιατί έχουμε καθυστερήσει. Ο κύριος Ντεσούτερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να απαντήσω σε τρεις παρατηρήσεις που έγιναν. Η πρώτη αφορά στο ερώτημα της κυρίας Μαγκίνες σχετικά με τα λάμπρες και τις προδιαγραφές που χρησιμοποιούν ε, οι μεγάλες ε, φίρμες ε, του εμπορίου. Πού ξεκινάει λοιπόν το λάμπελ, η επισήμανση και πού σταματάει η ανησυχία της επιχείρησης οι εταιρείε έχουν μία εικόνα που απορρέει και από τη διαφημίση και που ε, διασφαλίζει τον ε, <coughs> καταναλωτή. Η σήμανση δίνει εγγύηση βέβαια στον καταναλωτή και στην τιμή που θα πληρώσει. Εγώ να σας πω το εξή. Η οδηγία του 2005 για τις αφέμητες εμπορικές πρακτικές είναι η αναθεώρηση μιας οδηγίας του 1994 για την ε, παραπλανητική διαφήμιση. Θα μπορούσε να χρησιμοποιείται πολύ πιο συστηματικά για να καταπολεμούμε την ε, ψευδή διαφήμιση, τη διαφήμιση που οδηγεί σε λάχος. Δηλαδή αυτά τα ψευτολάμπελ τα οποία δεν αξίζουν για τίποτα. Και ακόμη και ο κώδικας συμπεριφοράς και αυτός θα πρέπει να ελέγχεται δηλαδή για, τη για την ψευδή διαφήμιση και οι φίρμες που χρησιμοποιούν αυτά τα labels, αυτή τη σήμανση που παγιδεύει τον καταναλωτή πρέπει να τιμωρηθούν. Οι νόμοι υπάρχουν. Θα πρέπει λοιπόν αυτοί που τους εφαρμόζουν να το κάνουν καλύτερα. Επίσης υπάρχει και ένα σημαντικός ρόλος που μπορεί να παιχτεί από την πληροφόρηση του καταναλωτή. Η σύγχυση είναι απόλυτη για τον καταναλωτή μεταξύ των διαφόρων λάμπελ που του προτείνονται. Γιατί Να Όταν λέμε εμείς αηφορία έχουμε μέσα προστασία του περιβάλλοντος, σεβασμό κοινωνικών ε, ε, μέτρων, ε, Πρέπει λοιπόν να δοθεί μια διευκρίνηση σε όλα αυτά, πρέπει να γίνουν καμπάνιες και επίσης να ετοιμάσουμε και τον καταναλωτή για την καταχρηστική χρήση αυτών των λάμπελ. Ο κύριος Ταραμπέλα ρώτησε κάτι σχετικά με τη... μίλησε μάλλον και είπε ότι η αστάθεια των τιμών αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα για τους παραγωγούς. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό το πρόβλημα μεγαλώνει συνεχώς. Λοιπόν, αυτή η αστάθεια έχει πολλούς ε, λόγους που γνωρίζουμε. Οι συμπεριφορές ε, των Γιωργών ανάλογα με το αν έχουν καλέσει κακές χρονιές που οδηγεί τελικά σε τεράστια πλεονάσματα ή σε ελλείμματα η ζήτηση και η εξέλιξη των τιμών στην αγορά, αλλά και νέα φαινόμενα. Η κερδοσκοπία για την οποία μιλήσαμε, αλλά και ένα θέμα για το οποίο δεν μιλήσαμε ακόμα, είναι η ενεργειακή εξάρτηση για την παραγωγή τροφίμων. Εμείς με τα αγροκαύσιμα σήμερα βλέπουμε να γίνεται μία συγχώνευση μεταξύ αγοράς τροφίμων και φυτοκαυσίμων. Επίσης η, α, η, βιο, η γεωργία εξαρτάται άμεσα από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, δηλαδή έχουμε πολλαπλασιάσει στη γεωργία κατά 20 την ε, εξάρτησή μας ε, για, στη χρήση των ορεικτών καυσίμων. Ναι, εμείς θα πρέπει να σταματήσουμε όλη τούτη την αστάθεια. Μπορούμε να το κάνουμε με την ε, χρήση των ε, τροφιμικών αποθεμάτων, με τον τρόπο που ανέφερε και ο κύριος Ταραμπέλα για, το στοκάζ, ε, για την αποθήκευση και, την, και τον στοκάζ. Και όταν έχουμε χαμηλές τιμές, το κράτος να αγοράζει αυτά τα αποθέματα. Επίσης, ο ρόλος της ΠΟΕ, το ανέφερε ο κύριος Ταραμπέλα, πρέπει να αλλάξουμε προσανατολισμό ριζικά. Η απολευθέρωση του παγκοσμίου εμπορίου συγκεντρώνει την παραγωγή με τις ορισμένες περιφέρειες και σε πιο ανταγωνιστικούς ε, παραγωγούς. Πρέπει να την αποκεντρώσουμε τη γεωργία, διότι ευνοούνται οι μεγαλοπαραγωγοί, κατά των μικροπαραγωγών οι οποίοι τελικά είναι αυτοί που παρέχουν και τη μεγαλύτερη κοινωνική υπηρεσία για την οποία δεν ανταμείβονται. Σήμερα και αυτό εγώ προσπαθώ να περάσω ως μήνυμα στην ΠΟΕ. Να ευνοήσουμε για την κάθε χώρα να αναπτύξει μέσα δημοσίων πολιτικών ρύθμισης της αγοράς ευελιξία. Πολλές φορές η ΠΟΕ δεν το, δεν το επιτρέπει αυτό και να ευνοήσει τη δυνατότητα αυτών των χωρών να έχουν τροφιμική ασφάλεια. Να ενισχύσει δηλαδή τους γεωργούς τους ε, προστατεύοντας τους από τον ντάμπινγκ και να προστατεύει και την ε, κουλτούρα, την αγροτική κουλτούρα αυτών των χωρών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κλάρκ. Ναι, συγγνώμη, δεν πρόλαβα να σημειώσω τα ονόματα όλων όσων ε, μίλησαν. Πολλοί αναφέρθηκαν στον Όμπουτσμαν ε, και στον κωδικά δικαιολογία. Όπω καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή, σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, το οικονομικό βήμα, το οικονομικό φόρουμ, σκεφτείτε περί της εισαγωγής κώδικα δεντολογίας ή όχι. Δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση, μπορεί να μην το πράξει, αλλά είναι υπό εξέλιξη η συζήτηση αυτή και όπως είπα, και στη δική μου παρέμβαση σε εθνικό επίπεδο στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζουμε να υπάρχει ένα ομπούτσμαν. Κάποιος αναφέρθηκε στο αν θα είναι εκούσιο ο χαρακτήρας ε, για τον κώδικα και αν θα υπάρχουν νομικά μέτρα που θα υποστηρίζουν τον κώδικα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία δεν επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε νομικά μέτρα αλλά να δώσουμε στον Ombudsman την εξουσία, την αρμοδιότητα να αποφασίσει ο ίδιος περί των διανέξεων. Έτσι λοιπόν είναι κάτι πολύ πιο ευέλικτο. Μιλάμε για ένα πιο ευέλικτο φορέα. Δεν χρειάζεται κάποιο να προσφύγει στα δικαστήρια. Ο Μπούτσμαν θα ακούσει τα αποδεικτικά στοιχεία και από τι δύο πλευρέ και θα έχει την εξουσία να αποφασίσει ποιο έχει δίκιο. Έτσι λοιπόν πρόκειται για μια ευέλικτη προσέγγιση. Αυτό είναι το θετικό. Επίσης, ε, κάποιοι έθεσαν την ερώτηση σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι να δούμε τι ισχύει για αυτό το τομέα, γιατί το άρθρο 82 Έχουμε το άρθρο 82 και βλέπουμε ότι επειδή τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν τεράστια μερίδια αγοράς ε, σε επίπεδο ένωσης, δεν ε, μιλάμε για μια παρόμοια κατάσταση όπως η Microsoft που μπορεί να κατέχει το 80% μιας συγκεκριμένη αγοράς. Δεν ε, βλέπουμε μια τέτοια κατάσταση στα τρόφιμα. Έτσι λοιπόν αυτό περιορίζει το πεδίο της Νομοθεσία περί ανταγωνισμού, δηλαδή ε, σε τέτοιες περιπτώσεις ε, θα ίσχυε για τις συγκεντρώσεις ε, στον τομέα των τροφίμων. Κάποιος είπε ότι θα πρέπει να περιορίσουμε το μέγεθο των ομιλών των σούπερ μάρκετ, όμως <laughs> Τίθεται ερώτηση και τι θα γίνει με τη Microsoft. Αν περιορίσετε το μέγεθο των ομίλων σούπερ μάρκετ, μπορεί να έχετε 15% τη αγορά Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι θα κάνετε με τη Microsoft που κατέχει το 80% του μεριδίου τη αγορά. Νομίζω ότι αυτά είναι προβλήματα που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού στον τομέα αυτό. Κάποιος αναφέρεται σε ιδιωτικές σημάνσεις. να σας πω ότι υπάρχουν και θετικά και αρνητικά ε, στι ιδιωτικέ σημάνσει, υπάρχουν και θετικά και αρνητικά στοιχεία. Το καλό είναι ότι μπορεί κάποιος να αγοράσει πιο φτηνό το προϊόν από ότι ε, θα αγοράσει ένα προϊόν που έχει ένα ισχυρό σήμα. Και κάτι ακόμα. Ο κύριος νομίζω Αναφέρθηκε στο αν υπάρχει δυνατότητα καλύτερης ρύθμισης στην αγορά, της αγοράς στον τομέα της γεωργίας. Είναι δύσκολο αυτό. Νομίζω ότι δεσμεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί προς ε, λιγότερη νομοθεσία στα πλαίσια της ε, ΚΑΠ. Εγώ το προτείνω για τον εξής λόγο. στα πλαίσια της ρύθμισης της αγοράς γάλακτος Λουχάρια. Τα πλεονεκτήματα το να θέσει κάποιος, ε, να καθορίσει κάποιος τιμές ε, είναι κάτι απλό. Έτσι λοιπόν ε, θα υπάρχει ο έλεγχος της τιμής, όμως φυσικά πρέπει να υπάρχει εκ των προτείνων σχεδιασμός και αν παράγεται πάρα πολύ γάλα, την επόμενη χρονιά θα μειώσετε την τιμή. Ε, όμως είναι απλή αυτή η διαδικασία. Όμως στις αγορές όπου υπάρχει και ποικιλομορφία στο εισόδημα, ίσως όχι στο γάλα, αλλά σε αγορές όπου αλλάζουν οι παράγοντες προσφοράς και ζήτησης, πρέπει να σκεφτείτε και τη σταθερότητα του εισοδήματο. Έτσι λοιπόν, ε, σε εκείνο το πλαίσιο, το να καθορίσει απλώς κάποιο μια τιμή δεν αρκεί. Θα πρέπει να λάβετε και μέτρα για τη σταθεροποίηση του εισοδήματο σε ορισμένους γεωργικούς τομείς. Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Ο κύριος Δηρία έχει το λόγο. Επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θα περιοριστώ σε τρεις ζητήματα και στο συγγνώμη από τους υπόλοιπους. Ε, κύριος Τραβέλα αναφερθήκε στο θέμα της αστάθειας. Καταρχήν, ε, νομίζω ότι εδώ μπορούμε να συμφωνήσουμε απόλυτα με τον κύριο Ντεσίτερ είναι κακή αστάθεια για όλους τους πρωταγωνιστές εκτός από τους κερδοσκόπους και πρέπει να ληφθούν μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Το δεύτερο θέμα που στο οποίο θέλω να φερθώ είναι το θέμα του Ombudsman. Είναι πραγματικά κάτι πολύ ενδιαφέρον. Συνήθως ε, οι Ombudsman, ε, οι διαμεσολαβητές υπερασπίζουν τους καταναλωτές και θα ήθελα να προτείνω να υπάρχει ένας διαμεσολαβητής μεταξύ των ε, λιανεμπόρων και των ε, ε, μεταποιητών που είναι οι μεγάλοι παίκτες. Ο κύριος Μποβέ έδωσε ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα της ε, αγοραστικής δύναμης που ασκείται έναντι των γεωργών καθηγητής ΛΑΙΑΝΣ που είναι αρμόδιος για ε, την εξέταση του θέματος της προσφοράς δεν υπόστηριξε ε, την αρχή ύπαρξης όμπουτσμαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και θέλω να πω ότι η ύπαρξη κωδικές διοντολογίας και τη μεσολογική εξαρτάται απόλυτα από την υφιστάμενη νομοθεσία. Εγώ θα αναφερθώ στην ιδέα που υποστήριξαν ε, κάποιοι ε, βουλευτές ότι η φυσταμένη νομοθεσία αρκεί, αλλά θα πρέπει να εφαρμοστεί καλύτερα από τη σήμερα. Και να προσθέσω ότι σχέση με το πιθανό διαμεσολαβητή στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο ε, κώδικας ε, δίνει ε, την δυνατότητα ε, τα μέρη να προσφύγουν σε αυθαίρετη επίλυση των διαφορών. Έτσι λοιπόν μπορεί να μην χρειάζεται ο Μπουτσμαν σε αυτή την περίπτωση, αλλά θα ήθελα να αφαιρθώ και στα σχόλια της κυρίας Γκίνες που είναι πολύ σημαντικά αναφέρθηκε στο θέμα της αγοραστικής ε, δύναμης ε, των λιανεμπόρων. Θα σας δώσω δύο νούμερα πολύ ε, μεγάλη λιανεμπόρη με βάση την Γαλλία. Ε, καταλαμβάνει το 30% ε, και εκπροσωπούν μόνο το 0,5% αυτού του ε, κατασκευαστή. Και στην Ισπανία, αν έχουν το 50% του μεριδίου της αγοράς, θα ήθελα να σας πω ότι οι κύριοι ε, τρεις παραγωγοί αναψυκτικών έχουν το 90% και οι πίτσες πρέπει το 70%. Έτσι λοιπόν το 50% είναι πολύ αλλά νομίζω το 70% είναι περισσότερο. Και νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι η ερώτηση της κυρίας Γκίνες για τις ιδιωτικές σημάνσεις και την πιθανή απαγόρευση αυτών ιδιωτικέ σημασίε δεν υπάρχουν κατά τύχη, αλλά ανταποκρίνονται στο αίτημα των καταναλωτών, δίνουν προστιθέμενη αξία, πιο καινοτόμα και φτηνότερα προϊόντα. Και θα ήθελα να πω ότι και οι μικρές και μισέ επιχειρήσει ε, τα θετούν. Αυτό ζητούμε σήμερα. Και ξέρετε ότι Μαρξ Σπέσερ ε, έχει το 99,9% της ειδικής σήμανσης ε, και εξακολουθούν να την προτιμούν οι καταναλωτές και αν δείτε ε, τι καταβάλλεται για το γάλα στους καταναλωτές θα σας πω ότι η Marks Spencer είναι η εταιρεία που πληρώνει τη δεύτερη ψηλότερη τιμή στους παραγωγούς. Έτσι λοιπόν μπορώ να σας πω ότι η ιδιωτική σήμανση μπορεί να είναι κάτι το οποίο αποφέρει κέρδος σε όλους τους εμπλεκομένους. Ευχαριστώ. Εδώ θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της ακρόασης. Θα περάσουμε τώρα στο δεύτερο μέρος και να ξεκινήσουμε με τον κύριο Φραντ Σίναμπελ του Αυστριακού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών, ο οποίος θα μας παρουσιάσει την άποψή του για το πώς η Ευρωπαϊκή Ελισίδια Εφοδιασμού Τροφίμων θα καταστεί πιο αηφόρος. Παρακαλώ. Uh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Το θέμα της ακροάσεως είναι δίκαιο εισόδημα για τους γεωργούς. Η ε, παρουσίασή μου <clears throat> θα έχει το ειδικότερο θέμα πώς να γίνει πιο ε, βιώσιμη η διατροφική, η αγροδιατροφική αλυσίδα. Ε, θα δείτε τα διάφορα θέματα που καθένας, κανένας θα μπορούσε να μιλήσει τουλάχιστον 10 λεπτά για καθένα από τα σημεία αυτά. Εγώ όμως θα ρίξω ιδιαίτερο βάρος στη, στο δίκαιο εισόδημα. Νομίζω ότι το δίκαιο εισόδημα έχει διαφορά από την δίκαιη τιμή. Πάντως η δίκαιη τιμή είναι ένα σημαντικό θέμα. Πρώτα θα ήθελα να ε, δώσω μια, έναν ορισμό εργασίας για την ε, ε, βιώσιμη ανάπτυξη, να κάνω ορισμένες σκέψεις σχετικά σε ορισμένες χώρες μέλη και μετά θα έρθω σε ορισμένες ε, επιλογές πολιτικής για να διευκολυνθεί η διατήρηση μιας βιώσιμης ανάπτυξης. Η ε, γεωργία παράγει τρόφιμα και ίνες. Ε, σημαντικά, αλλά όχι μόνο. Για παράδειγμα και άλλες παραγωγές μη αγαθών, δηλαδή για παράδειγμα υπηρεσίες οι υπηρεσίε από την αγροτική παραγωγή ανέρχονται σε 10 έως 15% σε ορισμένες χώρες μέλη και έχουμε και εκροές πολυλειτουργικές οι οποίες δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν μέσα στην αγροτική παραγωγή. Η, ε, η αγροτική παραγωγή επίσης αλλάζει στο ε, παρελθόν αυξανόταν διαρκώς η παραγωγικότητα της εργασίας. Τώρα διαπιστώνουμε ότι είναι χαμηλότερη σε πολλές ε, χώρες μέλη και βέβαια και το φαινόμενο αυτό είναι και παγκόσμιο. Θα έρθω τώρα ε, σε, μια, σε έναν μάλλον ορισμό της βιώσιμης ανάπτυξης στον χώρο της υπαίθρου. Ε, χρησιμοποιώ το μοντέλο ενός Ούγκρου οικονομολόγου, ο οποίος έχει φτιάξει μια πυραμίδα. Στην βάση της πυραμίδας αυτής ε, διαλαμβάνονται διάφορα στοιχεία που αποτελούν την βάση αυτού που θεωρούμε ότι είναι και ο αντικειμενικός σκοπός της ε, κοινωνίας. Αφενός το περιβάλλον. Είναι περιττό να πει κανεί ότι χρειάζεται ένα καλό περιβάλλον που να αποτελέσει τη βάση της γεωργίας. Και για να αποφευθούν ζημιές στο περιβάλλον χρειαζόμαστε ε, θεσμούς, κοινωνικούς θεσμούς οι οποίοι θα διευκολύνουν και την επίτευξη ε, Υψηλή παραγωγικότητας τη εργασία στη βάση ενός ε, καλού περιβάλλοντο Θα έρθω για λίγο τώρα στην παραγωγικότητα τη εργασία, η οποία αποτελεί κατά βάση συνάρτηση της εκπαίδευση, της παιδεία. Όσο πιο εκπαιδευμένοι είναι οι αγρότε, τόσο περισσότερες πιθανότητε έχουν να μπορούν να παράγουν ε, καλύτερα προϊόντα. Και βέβαια ο απότερο στόχο είναι βέβαια η ε, ποιότητα ζωής και ένα υψηλότερο βιωτικό επίπεδο. Υψηλότερο βιωτικό επίπεδο. Δεν μιλούμε μονάχα για χαμηλότερες τιμές. Οι χαμηλότερες τιμές συχνά σημαίνουν και χαμηλότερη ποιότητα. Ας έλθω τώρα στην ετερογένεια της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε σε πολλές χώρες μέλη οι γεωργοί να εργάζονται σε ε, περιοχές οι οποίες έχουν πυκνότερο πληθυσμό από άλλες ε, χώρες. Για παράδειγμα, στις κάτω χώρες, το Λουξεμβούργο και άλλες ε, χώρες που διαλαμβάνονται στην πρώτη ομάδα, η Οι γεωργοί μπορεί να έχουν και μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, όπως, είναι, όπως ε, συμβαίνει για παράδειγμα σε ορισμένε σκανδιναβικέ χώρε, αλλά είναι σε πολύ, στενό, ε, σε πολύ στενή διασύνδεση με τον καταναλωτή. Και αυτό είναι μια δυνατότητα υπέρ των παραγωγών να βελτιώσουν το εισόδημά του. Βλέπετε τώρα μια γραφική παράσταση. 500, 500 περίπου σημεία. Κάθε σημείο εκπροσωπεί μια περιοχή ΝΑΤΣ 3 ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. βλέπετε τα κιανά σημεία, δύο ε, απάνω δεξιά, στο δύο μάλλον απάνω δεξιά, όπου σημαίνει ότι υπήρξε σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια. Βλέπετε τώρα αριστερά περιοχές στην Ευρώπη όπου μειώνεται ο τομέας ε, της αγροτικής οικονομίας. Τώρα μιλούμε λοιπόν για δίκαιο εισόδημα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν περιοχές ή περιφέρειες που καθιστούν δυνατό να αυξάνουν το εισόδημά τους οι γεωργοί, κυρίως όπου οι οικονομίες συνολικότερα αναπτύσσονται καλύτερα. Οι συνέπειες τώρα. Νομίζω ότι η εγχώρια πολιτική ανταγωνισμού παίζει σημαντικό ρόλο. Γνωρίζομαι ότι οι πολιτικές ανταγωνισμού διαμορφώνονται διαφορετικά στις διάφορες χώρες μέλη. Βασικός στόχος τους είναι βέβαια να ωφελήσουν τον καταναλωτή. Οι τιμές θα πρέπει να είναι χαμηλές, όχι όμως πάρα πολύ χαμηλέ, χαμηλές, ώστε να αποτρέπεται η αύξηση της ποιότητας και η καινοτομία. Εγώ προέρχομαι από την Κεντρική Ευρώπη. Νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε πολλά πράγματα από την πολιτική ανταγωνισμού που ασκείται στο Ενωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία. Αλλά μπορούμε να κοιτάξουμε και λίγο πιο μακριά στις Ενωμένες Πολιτείες, όπου βλέπουμε ότι η πολιτική ανταγωνισμού είναι θέμα που έχουν πάρει στα χέρια τους καταναλωτές και έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στα δικαστήρια. Και έτσι οι καταναλωτές μπορούν να εξαναγκάσουν παραγωγούς και ηλιανικό εμπόριο να απόσχουν από ε, συμπεριφορά που βλάπτει τον ανταγωνισμό. Πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν τον καταναλωτή μέσα στην, ε, στο πλαίσιο αυτού του ανταγωνισμού. Η παραγωγή βέβαια χρειάζονται ομαλό πεδίο ανταγωνισμού. Επίσης το διεθνές εμπόριο είναι σημαντικό, διότι οι, οι παραγωγοί έχουν ανάγκη να έχουν πρόσβαση σε πόρους και διεθνώς και οι ε, καταναλωτές πρέπει να έχουν υψηλό εισόδημα για να μπορούν να καταναλώνουν τα προϊόντα, τα αγροτικά προϊόντα. Η καινοτομία και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Άλλη λοιπόν πολιτική επιλογή. Μάλλον πολιτική επιλογή. Αγροτικές πολιτικές που ε, δίνουν ιδιαίτερο πάρος στις επενδύσεις. Βλέπουμε να σημειώνεται μια ε, σχετική μείωση, παρακμή της αγροτικής έρευνας και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στις Ενωμένες Πολιτείες. Γνωρίζουμε ότι για δεκαετίες οι καταναλωτές επωφελήθηκαν από χαμηλότερες τιμές. Όχι επειδή το ελληνικό εμπόριο ήταν τόσο ανταγωνιστικό ώστε να μειώνονται οι τιμές, αλλά επειδή υπήρξαν τεράστιες επενδύσεις, δημόσιες επενδύσεις στην έρευνα, ώστε η αγροτική εκμετάλλευση να γίνει πιο παραγωγική και να αυξηθεί το παραγόμενο προϊόν. Βλέπουμε τώρα να μειώνονται οι επενδύσεις αυτές. Μία από τις συνέπειες θα είναι οι τιμές ενδεχομένως να αυξηθούν στο μέλλον. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε την τεχνολογία ούτω ώστε να είναι βιώσιμη η ανάπτυξη γιατί γνωρίζουμε ότι νέες τεχνολογίες αποτελούν προϋπόθεση για μείωση των βλαβών του περιβάλλοντος. Και νομίζω ότι τουλάχιστον σε ορισμένες χώρες μέλη χρειαζόμαστε και καλύτερη καλύτερες διαδικασίες για την επίλυση διαφορών. Και θα τελειώσω με την διαφάνεια που ε, δείχνω τώρα, που δείχνει την διασύνδεση μεταξύ των τιμών των ορυκτών καυσίμων, αριστερά, στην κάθετο δηλαδή, και τιμές του σταριού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει σαφής διασύνδεση. Όσο αυξάνει η τιμή του ορυκτού καυσίμου, τόσο αυξάνει και η τιμή του ΣΥΤΟΥ. Εδώ μπορούν να παίξουν ένα ρόλο και αυτοί που αποφασίζουν ποιες επενδύσεις θα γίνουν στην ε, δημόσια επενδύση, δηλαδή θα γίνουν στην έρευνα για γεωργικά προϊόντα και με τον τρόπο αυτό μπορούν να επηρεάσουν την καμπύλη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φραντσέσκο Κόντο, καθηγητής της οικονομίας στο Πανεπιστήμιο της Φότζα. για τα ωφέλη για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές στα πλαίσια μιας αυξημένης ανταγωνιστικότητας. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ αφού πω ότι συμφωνώ το μάλλον με την έκθεση του κ. Μποβέ, θα ήθελα να συνεισφέρω στη συζήτηση αυτή με μια μεθοδολογική προσέγγιση διαφορετική. Θα ήθελα να εισαγάγω τους ε, εξωτερικούς ε, παράγοντες ε, στην αγροτροφική λυσίδα αυτή καθ' αυτή. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Εμείς ε, έχουμε εδώ μία σύνθεση της κλασικής διατροφικής αλυσίδας που αποτελείται από τους γεωργούς, τους χονδρέμπορους, τους ενδιάμεσους και τους και έχουμε την ε, διανομή και το γενικό τομέα. Όλοι αυτοί οι πρωταγωνιστές, ε, αν θεωρηθούν ως ένα και μόνο οικονομικό υποκείμενο, αυτό που λέμε εμείς ο τομέας, έχουν με τη σειρά τους οικονομικές σχέσεις με εξωτερικούς ε, πρωταγωνιστές και θα αναφέρω ε, σε ποιους εμείς επικεντρωνόμαστε στην ομάδα μελέτης στην Ιταλία. Ενδιαφερόμαστε στις επιχειρήσεις επικοινωνίας και πρόθεσης, ε, τους ε, ε, προμηθευτές εφοδιαστικής, τους προμηθευτές ενέργειας και ακούσαμε αναφορές σε αυτούς, τους προμηθευτές συσκευασία τεχνικών μέσων για τη γεωργία, προμηθευτές πρόσθετων ουσιών, τεχνολογίας και υπηρεσιών συμβουλευτικών στη γεωργία. Αν ε, εμείς δούμε όπως ε, κάναμε σε πρόσφατες και σβάθος ε, μικροοικονομικές μελέτες στην Ιταλία, συνειδητοποιούμε ότι το εσωτερικό κόστος στον γεωπιστητικό τομέα αυτό καθευτό φτάνουν στο να ε, δημιουργούν στο να φτάνουν στο 3% σε χρήσιμη παραγωγή. Αυτό το 3% το μοιράζεται η γεωργία. Ε, δηλαδή ας φανταστούμε 3 ευρώ. Και αν μιλήσουμε για 3 ευρώ έχουμε 70 λεπτά ε, για τη βιομηχανία, 30 ε, η μεταφορά 0,40 ε, η τροφοδοσία ενώ τα υπόλοιπα καλύπτουν εσωτερικό κόστος του τομέα και έχουμε 38% κόστος εργασίας, 11% κόστος κεφαλαίου που κυρίως δημιουργείται από τις εξοφλήσεις και από τα επενδυτικά αγαθά και 5% το κόστος ε, χρηματοδότησης. Κυρίως αναφέρομαι στις ε, προμήθειες που λαμβάνουν οι τράπεζες και έχουμε και 27 ευρώ στο 100 τα οποία δίνονται και Θέλω να επικεντρωθώ αυτό. Έχουμε 8,5 ευρώ στη συσκευασία, 5 ε, ευρώ στη μεταφορά, 5 ευρώ σε όλες τις δραστηριότητες προώθησης, 3,7 ευρώ στην ενέργεια, 1,20 στα τεχνικά μέσα και 2,9 ευρώ σε μια σειρά άλλων υπηρεσιών. Και κατόπιν, για να συμπληρώσουμε, έχουμε 12 ευρώ για τους φόρους και ε, έχουμε και 0,25 που αφορούν τις, μάλλον το 1 τέταρτο, με συγχωρείτε, εισαγωγές από το εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν σας ρωτήσω κύριε Μποβέ είναι πράγματι ιδιαίτερα παραγωγικό για τη συλλογιστική μας αν ο στόχος μας είναι να έχουμε πιο υψηλές οδήματα για τους γεωργούς να αναλαμβάνουμε δράσεις για να αφαιρέσουμε εισόδημα από άλλους πρωταγωνιστές στο εσωτερικό τομέα. Δηλαδή, δεδομένου ότου μιλάμε για ένα τόσο μικρό ποσό, 3 ευρώ στα 100 σε συνολικές δαπάνες. Και όπως υπόθηκε στην αρχή να σας πω ότι εγώ συμφωνώ όταν μιλάμε μόνο για τον τομέα στο εσωτερικό του. Ε, συμφωνώ με τις ε, ενδείξεις που δίνεται στην έκθεση, όμως εγώ θεωρώ ότι είναι πιο χρήσιμο να επανέλθω σε αυτά τα θέματα στο τέλος. Θεωρώ πιο χρήσιμο να επικεντρωθώ στο εξή. Το αν εμεί θέλουμε τώρα να αυξήσουμε το εισόδημα των γεωργών και να δράσουμε έτσι ώστε η Επιτροπή Γεωργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να είναι πιο αποφασιστική επί μια σειρά ε, επιχειρημάτων που θα εθετήσει, που θα αναφέρω τώρα και αυτή θα είναι και η συνεισφορά που θέλω να κάνω εγώ σε αυτή τη συζήτηση το να μειώσουμε το εργασιακό κόστος, ε, το εργασιακό κόστος κυρίως για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ε, αλλά και για τους ε, άλλους εσωτερικούς πρωταγωνιστές του τομέα. Το να συγκρατήσουμε το εξωτερικό κόστος του τομέα είναι ένα θέμα κεντρικό εξωτερικό κόστος όπως είναι οι μεταφορές, η εφοδιαστική, η συσκευασία, η ενέργεια και τα τεχνικά μέσα επί των οποίων αναφέρθηκαν και άλλοι συνάδελφοι. Να ε, δεσμεύσουμε μέσω μιας δράσης ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα κράτη να μειώσουν ε, τους φόρους και το κόστος της ασφάλισης. Ε, στη συνέχεια να μειώσουν το γραφειοκρατικό κόστος ε, που έχουν σημαντική επίπτωση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στους υπόλοιπους πρωταγωνιστές τομέα και να περιορίσουν τις εισαγωγές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ευνοήσουν αντίθετα την εργοποίηση του πράσινου διαδρόμου κυρίως για τις παραγωγές από τις μεσογειακές χώρες. Και θα κάνω κάποιες προτάσεις για κάθε ένα από τα σημεία αυτά. Πώς θα μειώσουμε το κόστος εργασίας να επιβεβαιώσουμε διευκολύνσεις για ορισμένες ε, ορεινές περιοχές, ε, να μειώσουμε τους ε, φόρους για την πρόσληψη εργατικού δυναμικού, δηλαδή να ευνοήσουμε όλους τους εργοδότες οι οποίοι προσφέρουν πολλές θέσεις εργασίας ή διασφαλίζουν ότι θα προσφέρουν πολλές ημέρες εργασίας. Πώς θα μειώσουμε τώρα το εξωτερικό κόστος του γεπιστικού τομέα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να δώσουν κίνητρα στα κράτη έτσι ώστε να μπορέσουν να συνάψουν συμβάσεις με ε, πιο χαμηλό κόστος για τις ε, διεθνείς αποστολές για το πιστιστικό προϊόντων να ε, υλοποιήσουν μια συγκεκριμένη πολιτική δημόσιας παρέμβαση για να βελτιώσουν τις υποδομές για την ε, εφοδιαστική του τομέα και θα σας πω ένα παράδειγμα να είναι υποχρεωτικό ένα ποσοστό επενδύσεων από τα κράτη-μέλη υπέρ αυτής της υποδομής στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΦΕΣΡ γιατί ξέρετε ότι όταν το ΦΕΣΡ εισήχθη οι περιφερειές μας και τα κράτη μας ε, τώρα ε, έχουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα της ανάπτυξης της υπαίθρου, της αγροτικής ανάπτυξης και ε, οι ε, πτυχές τι, του της γεωργίας αποκλείονται, ενώ οι πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται για άλλους τομείς. Και εγώ νομίζω ότι αυτοί οι πόροι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ε, στο γεωπεσητιστικό τομέα και στις σχετικές υποδομές. Θα μπορούσαμε επίσης να ε, έχουμε μεγαλύτερες επενδύσεις ε, στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, αιωλική, φωτοβολταϊκή κτλ. Γιατί αποτελούν και εναλλακτική πηγή εισοδήματος για τους παραγωγούς, αλλά μπορούν και να μειώσουν το κόστος της ενέργειας μπορούμε να εξαλείψουμε τα διάφορα ε, περιβαλλοντικά εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν στην νομοθεσία των κρατών μελών. Επίσης, να προωθήσουμε κοινοτικέ πολιτικές που ευνοούν την απελευθέρωση της αγοράς των τεχνικών μέσων και τη δημιουργία ομάδων ε, συλλογικών αγορών. Ξέρουμε πόσο ε, οι πολυεθνικές, πόσο μεγάλο ρόλο διαδραματίζουν οι πολυεθνικές σε αυτό το θέμα των τεχνικών μέσων. Επίσης, ε, να δοθεί ανατολισμό στα κράτη να μειώσουν τους φόρους, το ΦΠΑ, ε, λόγου χάρη και κάτι τέτοιο θα διευκόλυνε και τους καταναλωτές, αλλά θα ευνοούσε και την αύξηση της κατανάλωσης και την αύξηση του εισοδήματο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης επί των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, μείωση των ε, άμεσων φόρων σε συγκεκριμένους τομείς. Και εμείς προτείνουμε ε, ένα είδος ελεύθερης ζώνης ε, για ε, τα ποιοτικά προϊόντα και για συγκεκριμένους παραγωγικούς τομείς που σε συγκεκριμένες, πτυχές, σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές θα μπορούσαν να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα. Πώς να μειώσουμε τώρα το κόστος της γραφειοκρατίας, νομοθετική απλούστευση σε περιφερειακό εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ένωσης. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πληροφορική για το σκοπό αυτό και τις νέες τεχνολογίες πώς θα περιορίσουμε ε, τις εισαγωγές ε, από τρίτες χώρες, ε, να μειώσουμε το ποσοστό των πρώτων υλών που εισάγονται και μεταποιούνται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια πρακτική ιδιαίτερα συνήθις δυστυχώς, να εγγυθούμε πραγματική ρύθμιση των τιμών των πρώτων υλών στον τομέα της γεωργίας, να σεβόμαστε περισσότερο του ε, υγειονομικούς κανόνες από τις τρίτες χώρες. Και ας έλθουμε τώρα στις πολιτικές που θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει εφαρμογή κατά την άποψή μα για να βελτιώσει το εισόδημα των γεωργών μέσω μια πιο αποτελεσματική λειτουργία ε, του γεωπιστικού τομέα. Και μέσω μιας καλύτερης ρύθμισης ε, των πιστοποιητικών ποιότητας. Ε, επιλαμβάνω ότι αναφέρομαι σε αυτή τη μεθοδολογική προσέγγιση που αφορά εξωτερικούς ε, παράγοντες του τομέα για τους λόγους που εμείς θεωρούμε σημαντικούς γιατί θα μπορούσαν να συμβάλλουν στο να αυξηθεί το εισόδημα του Γεωργού. Θα ήθελα όμως τώρα να αναφερθώ στο εσωτερικό σκέλος του τομέα. Ε, να φέρουμε κάποιες προτάσεις που αφορούν τέσσερις τομείς παρέμβασης. Ε, παρέμβαση για την ενθάρρυνση των συμφωνιών ε, στον τομέα, να δοθούν κονδύλια για την τεχνολογική έρευνα προς την πραγματική εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Γεωργών, να ρυθμιστούν με διαφορετικό τρόπο οι πολιτικές παρέμβασεις που υλοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την, τον λεγόμενο ευρύ τομέα από αυτές για το λεγόμενο πιο περιορισμένο τομέα να ε, εξεταστεί εκ νέου το σύστημα πιστοποίησης ποιότητας. Σας έρθουμε στο πρώτο. Έχουμε παρεμβάσεις για τη διευκολύνση των συμφωνιών. Ξέρετε ότι ο τομέας δεν ε, είναι κάτι που συναντάμε σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρομαι κυρίως ε, στις χώρες της ε, νέας, τις νέες χώρες και σε χώρες της Μεσογείου. Αυτό έχει γίνει μέσω των PSR, μέσω των ε, σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να παραχθεί προστασία στους γεωργούς από το να τους εκμεταλλεύονται κάποιοι άλλοι πρωταγωνιστές του τομέα. Μιλήσατε για δεσπόζουσα θέση. Εγώ συμφωνώ με τις ε, παρεμβάσεις σας, αλλά νομίζω ότι μπορούν να γίνουν και περισσότερα. Να προωθήσουμε τις ε, οργανώσεις προϊόντων και όχι μόνο οργανώσεις παραγωγών, διευρύνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτές τις οργανώσεις προϊόντος ε, σε αυτές να μπορούν να συμμετέχουν και ε, μη γεωργοί. Ε, επίσης, θα πρέπει μέσω της νομοθεσίας να αναθεωρούμε και αυτά τα περιφερειακά προγράμματα και τα ολοκληρωμένα προγράμματα του τομέα. Για την έρευνα, αναδιάρθρωση Ε, το τρόπο που υλοποιούνται οι διαγωνισμοί για να χρησιμοποιηθούν καλύτερα οι πόροι που προβλέπονται από τα εθνικά προγράμματα για την έρευνα υπέρ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που σήμερα δυστυχώς ε, διέπονται από συμφέροντα Ινστιτούτων Έρευνας και Πανεπιστημίων. Η έρευνα ε, θα πρέπει να, είναι, να χρησιμεύει για τη βελτίωση της ποιότητας. Τώρα, για τους δύο τομείς, τον ευρύ τομέα και τον πιο περιορισμένο τομέα. Εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω μια συγκεκριμένη πτυχή ε, του πιο περιορισμένου τομέα. Δηλαδή, τομεί στου προστατευμένου τομεί. Α μιλήσουμε για του μικρού παραγωγού. Ε, έχουμε κάποιου τομεί ε, οι οποίοι θα πρέπει να επικεντρώνουν στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και θα πρέπει να έχουμε και κάποιους τομείς εγκύτητας, δηλαδή οι μικροί παραγωγοί να έρχονται πιο κοντά στην τοπική αγορά και να γίνεται συγκεκριμένη αναφορά και στις τουριστικές δραστηριότητες. Και επίσης παρεμβάσεις υπέρ τη ποιότητα, το να επιλεχθεί ένα κατάλογο προϊόντων αριστείας σε κοινοτικό επίπεδο ε, και να δίνονται σε αυτά συγκεκριμένε σημάνσεις και να αναγνωρίζονται και στον ΠΟΕ υποχρέωση ένδειξης προέλευσης της πρώτης γεωργικής ύλης στην ετικέτα, ε, να δημιουργηθεί ειδικό ταμείο στο πλαίσιο του ΦΕΣ για να προστατεύονται αυτά τα προϊόντα από την παραποίηση και να παρέχεται και νομική αρρωγή στο εσωτερικό και στους ε, διεθνείς αγορές να προωθούνται αυτά τα προϊόντα. Επίσης, πολέμηση της παραποίησης και υποστήριξη των τιμών ε, σε επίπεδο ε, εκμετάλλευσης, να μειωθεί το κόστος υπέρ των γεωργών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, καθηγητά. Ο Πέδρο Πιμεντέλ, Γενικός Γραμματέας της Πορτογαλικής ΓΕΣΕ. Θα μας προτείνει λύσεις ώστε οι γαλακτοπαραγωγοί να έχουν πιο δίκαιες τιμές. Και θα μας μιλήσει και για τα δίκαια συμβόλαια στην αγορά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να σας πω ε, ορισμένα στοιχεία για την γαλακτοκομικό τομέα στην Πορτογαλία. Μου ζητήσατε όμως ε, να είμαι πολύ σύντομος, επομένως ε, θα το πράξω. Θα ήθελα να σας πω ότι η παρέμβασή μου είναι προσωπικού χαρακτήρα και δεν θέλω να δεσμεύσω τον πορτογαλικό, το γαλακτοκομικό τομέα. ο τομέας ο γαλακτοκομικός αναπτύσσεται με διάφορες μορφές στα κράτη με μελη Εν τω μεταξύ, παρόλα αυτά, θα ήθελα να απαντήσω στα δύο ερωτήματα που μου θέσατε. Πώ να διασφαλίσουμε ότι η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων μπορεί να χαίρουν δίκαιο τιμό στην λυσίδη των τροφίμων και αν θα είναι δυνατόν να υπάρχουν δικέ συμβάσει μεταξύ των μερών. Τι εννοούμε δικέ τιμέ, Πρέπει να υπενθυμίσω ότι αυτή η τιμή ισχύει και για τον παραγωγό αλλά και για όλου του άλλου πρωταγωνιστές της αλυσίδα. Εδώ πρέπει να μιλάμε και για μια σταθερή τιμή, όσο το δυνατόν πιο σταθερή να είναι ε, η τιμή αυτή. Επίση πρέπει να δούμε τι εννοούμε όταν μιλάμε για αστάθεια των τιμών. Αυτή η αστάθεια προκύπτει όταν υπάρχουν ενισορροπίες μεταξύ προσφορά και ζήτηση στην αγορά. Εμεί θεωρούμε θα πρέπει να υπάρχει υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά στην αγορά αυτή από ό,τι στις χρηματοοικονομικές αγορές και ε, φυσικά αυτές οι αστάθειες οφείλονται στην απορρίθμιση αυτών των ίδιων αγορών και στον ρόλο των κερδοσκόπων. Η απορρίθμιση της αγοράς και η διάλυση του σύμμεστος των ποσοστώσεων αυξάνει ε, τον κίνδυνο της αστάθειας ε, των τιμών και αυτό φυσικά δυσκολεύει τους παραγωγούς αλλά και την ίδια τη βιομηχανία. Η ίδια απορρίθμιση των αγορών φέρει και άλλη μια συνέπεια την αστάθεια των παραγόμενων ποσοτήτων ε, και φυσικά εδώ είχαμε τη φιλοσοφία των ποσοστώσεων και Εκεί τίθεται το κύριο θέμα ότι έχουμε ασταθείς όγκους παραγωγής γάλακτος ποτέ ε, στο γαλακτοκομικό τομέα δεν έλειψαν να υπάρχουν ε, τα προβλήματα ακόμη και όταν υπήρχε το, ποσοστό, το σύστημα των ποσοστώσεων. Είναι μια κοινή πρακτική. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχει σύναψη συμβάσεων στον τομέα, όμως υπό το καθεστώς των ποσοστώσεων αυτές οι συμβάσεις ρύθμιζαν τη διαδικασία μεταξύ των, των μερών και ε, στο πλαίσιο της λειτουργίας της αγοράς ήθελαν να ε, καταρτήσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και των δύο μερών. Αυτές οι συμβάσεις ε, δεν επιζητούσαν τη ρύθμιση των αγορών ή να ρυθμίσουν την προσφορά όταν βλέπουμε σήμερα ε, τι μπορούν να προσφέρουν οι συμβάσεις. Είναι ένα μέσο για να καταπολεμήσουμε την υπερβολική αστάθεια. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για συμβάσεις που συστήνεται με άλλη φιλοσοφία. Μιλήσουμε για, αν μιλάμε για αστάθεια, την υπερβολική αστάθεια, ε, μπορούμε να εμπνευστούμε από καταστάσεις που είδαμε στο παρελθόν ότι, υπήρξαν μαζική, ότι μαζική παραγωγή και δεν μπορούσε ξαναρυθμιστεί να χωρίς να υπάρχει εξωτερική παρέμβαση και είδαμε σημαντική μείωση στα εισοδήματα. Αλλά επίσης μπορώ να σας ε, περιγράψω και άλλες περιπτώσεις ε, είδαμε ότι αυτή η αστάθεια ήταν ε, στο ανώτερο επίπεδο της καμπύλης των τιμών. Το είδαμε το 2007 πέρα από όλη αυτή την κατάσταση με τους κύκλους και τους αντικύκλους. Εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες διαφορές σε σχέση με το πώς εξελίσσονται οι κύκλοι αυτοί όταν ε, η βιομηχανία δεν έχει ε, όγκους ε, παραγωγής για τη μεταποίηση, τότε υπάρχουν αντιδράσεις στον τομέα, διαφορετικές αντιδράσεις από ότι αν ο τομέας ακολουθούσε την κανονική κυκλική διαδικασία. Υπάρχουν κάποιες εκμεταλλεύσεις οι οποίες, ε, μάλλον συγγνώμη, βλέπουμε ότι πολλές φορές εισάγονται στην αγορά υπερβολική ε, όγκη παραγωγής ε, γάλακτος. Όταν ε, έχουμε τέτοιες περιπτώσεις η πιο λογική αντίδραση είναι να προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε το από θέματα να μειώσουμε την παραγωγή και να προσπαθήσουμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτηση, όμως η γαλακτοκομική παραγωγή γίνεται σε χιλιάδες εκμεταλλεύσεις και ε, κάθε παραγωγός δεν ε, έχει την ικανότητα να έχει ε, ικανή ένταξη στην αγορά για να μπορέσει να ρυθμίσει το πόσο λειτουργεί η αγορά και πρέπει να δούμε αν η τιμή που δίνεται είναι συμβατή με το κόστος παραγωγής και Πρέπει να δούμε αν έχουμε περισσότερη παραγωγή, αν αυτό σημαίνει και μεγαλύτερο εισόδημα για τον παραγωγό. Έχουμε όμως και άλλους παράγοντες που ρυθμίζουν στην αγορά, όπως τους διοικητικούς παράγοντες και υπάρχουν τεράστιες γραφειοκρατικές δυσκολίες. Όλες αυτές οι διαπιστώσεις αναφέρονται ε, το, μάλλον όλες αυτές τις δυσκολίες έλαβαν χώρα ε, παρά την ε, ύπαρξη του συστήματος ε, των ποσοστώσεων. Όμως πάντοτε πρέπει να έχουμε ελεύθερη έκφραση της βούλησης μεταξύ των δύο μερών και πρέπει να γίνεται σεβαστή, σεβαστός ο ανταγωνισμός. Ε, κατά τη γνώμη μου, ε, αυτές ε, οι συμβάσεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν ένα εργαλείο για να αποτραπεί η υπερβολική αστάθεια των τιμών στην αγορά. Το σύστημα των ποσοστάσεων μας οδηγεί και σε μια καλύτερη ανάλυση της αγοράς. Μία από τις πτυχές που προκύπτει από το καθεστώς ε, αυτό ε, της, της απώλειας του καθεστώτος των ποσοστώσεων είναι ότι δεν έχουμε πλέον τις κατάλληλες πληροφορίες. Δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της αγοράς. Και ε, Τώρα, πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτή τη σχολεία, να καθαστήσουμε υποχρεωτικές αυτές τις συμβάσεις, να εναρμονίσουμε το περιεχόμενό τους, να έχουν ένα δημόσιο χαρακτήρα, να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση και να έχουμε ένα έγγραφο στο οποίο θα καταγράφεται η ελεύθερη βούληση και των δύο μερών εκείνη τη στιγμή. Ε, στα διάφορα κράτη-μέλη βλέπουμε όμως ότι τώρα ακολουθούνται διαφορετικά μοντέλα. Θα έπρεπε να έχουμε ένα μοντέλο που να ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ισχύει σε όλη την κοινοτική επικράτεια. Όταν μιλάμε για ρύθμιση, ε, πάντοτε θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την παραγωγή και τη ζήτηση θα πρέπει να έχουμε υπόψη τους όγκους που υπάρχουν στην αγορά. Αν ε, θέλουμε να περιορίσουμε, πώς θα μπορούμε να περιορίσουμε τη ροή όταν έχουμε εντελώς ανομοιογενείς επιχειρήσεις στην αγορά, όταν έχουμε τελείως ε, ανομοιογενή γεωγραφική κάλυψη και από την άλλη ο ίδιος ο παραγωγός δεν μπορεί να καθορίσει ε, να έχει επίδραση στην αγορά. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε και την περίοδο της αστάθειας που έλαβε χώρα. Θα πρέπει να δούμε τι παράγεται από κάθε εκμετάλλευση και να δούμε αν για κάθε εκμετάλλευση πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη ποσόστοση παραγωγής. Ο παραγωγός αντιμετωπίζει διάφορες δυσκολίες ε, κατά την παραγωγή και ε, αυτός ε, πρέπει να ξέρετε ότι παράγει, ε, όμως αντιμετωπίζει διάφορους αστάθμιτους παράγοντες. Μπορούμε παραδείγματο χάρη να έχουμε προβλήματα που προκύπτουν από τις κλιματικές αλλαγές ή στην υγεία των ζώων. Το αν θα έχει ικανότητα να θέσει σε εμπορία ε, το, τις ποσότητες του γάλακτος για τις οποίες έχει, συμβα... έχει υπογράψει σύμβαση, αυτό θα πρέπει να το δούμε αν μπορεί να το πράξει. Και επίσης αυτές είναι αρισμονισμένες συμβάσεις πρέπει να ε, ρυθμίζουν την προμήθεια για μια διευρυμένη περίοδο ε, χρονική μία δίκαιη τιμή, θα πρέπει να καλύπτει το κόστος της παραγωγής, θα πρέπει να καλύπτει ε, το κόστος της εργασίας και θα πρέπει και να καλύπτει και τον κίνδυνο της επένδυσης. Αυτό είναι σχετικό για όλους τους κρίκους της ε, αλυσίδας. Επίσης ε, θα πρέπει να δούμε αν οι ανταγωνιστικές δυνάμεις της αγοράς είναι αυτές που καθορίζουν την τιμή της πώληση και όλη η δομή στη συνέχεια ε, χρησιμοποιείται για να καθορίσει και την τιμή του προϊόντος στο ράφι. Ε, δεν πρέπει ποτέ ένα προϊόν να απολύεται κάτω από το κόστος παραγωγής του και ε, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη πάντοτε τις ανταγωνιστικές δυνάμεις που υπάρχουν σε μια συγκεκριμένη αγορά. Επίσης, ε, πρέπει να κάνουμε και μια διάκριση μεταξύ των επιχειρήσεων ε, σήμερα. Βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο καταστάσεις όπου έχουμε πολύ διαφορετικές τιμές στα ράφια, ενώ η τιμή που πληρώνεται στο παραγωγό είναι η ίδια. Δηλαδή αυξάνεται το κόστος, αλλά δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία. Ε, ε, θα ε, έπρεπε τελικά να χρησιμοποιηθούν με καλό τρόπο οι πληροφορίες. Όταν η πολιτική συζήτηση επικεντρώνεται στο να δοθεί μια, ένα δίκαιο εισόδημα στο παραγωγό και όταν η συζήτηση αυτή τίθεται μόνο σε σχέση ε, με το παραγωγό και τη βιομηχανία, σαν να βρισκόμαστε σε ένα απομονωμένο κόσμο, ε, εγώ νομίζω ότι τελικά βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Γιατί ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη συνολική εικόνα του τομέα, γιατί διαφορετικά πολύ δύσκολα θα δοθεί ένα δίκαιο εισόδημα στον παραγωγό. Πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη και ποια είναι η τιμή που πληρώνει και ο καταναλωτής ε, αν θέλουμε να επιλύσουμε αυτές τις δυσκολίες, ε, τότε πάντοτε θα είναι δυνατό να πληρώνουμε ένα καλύτερο εισόδημα για τον παραγωγό. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Τελειώσαμε με τους εμπειρογνώμους. Όχι, όχι, έχουμε ακόμη έναν. Τον τελευταίο έχουμε τώρα. Λοιπόν, από το Βρόκλαβ ο κύριος Κοβάλσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί βουλευτές, σας ευχαριστώ όλους για την δυνατότητα που μου δίνεται να τοποθετούμε σήμερα στην Επιτροπή Γεωργίας. Το θέμα αφορά στα κριτήρια για την βιομηχανία τροφίμων, της βιομηχανίας τροφίμων προς τους αγρότες. Πρώτη παρατήρηση. Υπάρχει ένα, ε, ε, ένας κυρίαρχος κρίκος ε, της αλυσίδας Σήμερα θα μπορούσε, ε, μιλάμε σήμερα για την αγροδιατροφική αλυσίδα, δεν είναι ε, εδώ ο τόπος και ο χρόνος για να συζητήσουμε τις διαφορές μεταξύ αγροτικής βιομηχανίας και ε, διατροφικής αλυσίδας. Πάντως, στην ιστορία μέχρι τώρα υπήρχαν διαφορετικοί κρίκοι της αλυσίδας, της αγροδιατροφικής αλυσίδας, που ήταν κυριαρχή. Δηλαδή, επίκυλε αυτό, περνούσαν από τον ακρικό στον άλλο. και αυτοί οι κρίκοι υπαγόρευσαν τους τρόπους λειτουργίας της διατροφικής αλυσίδας. Ήταν ε, ο τομέας ε, της ε, προσφοράς στις δεκαετίες 40 και 50, μετά ήταν ο τομέας της μεταποίησης στις δεκαετίες 60 και 80, επειδή τότε η λιανική διανομή δεν ήταν τόσο εξελιγμένη και τώρα το λιανικό εμπόριο από τη δεκαετία του 80 και μέχρι και σήμερα. Με μια επιφύλαξη ότι δεν είναι βέβαια ακριβή τα χρονικά αυτά όρια. Χρειάζονται βέβαια και προσαρμογές αναλόγως με τις περιφέρειες ή τις ε, χώρες. Πάντως, από ό,τι βλέπετε, η ε, παραγωγή, οι αγρότες δηλαδή, ποτέ δεν ήταν ο κυρίαρχος κρίκος. Και αυτό καθορίζει τη δύναμη των ε, παραγωγών. Και γι' αυτό συζητούμε σήμερα το εισόδημα των ε, ε, αγροτικών παραγωγών και όχι το εισόδημα των μεταποιητών ή των διακινητών, του λιανικού εμπορίου δηλαδή. Αυτά είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Η δεύτερη τώρα παρατήρηση μπαίνει ως ερώτηση. Γιατί η βιομηχανία παραγωγής τροφίμου έχει τη δυνατότητα να απαιτεί διάφορα πράγματα από τους ε, ε, αγροτικούς παραγωγούς σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων. Προέρχεται αυτή η δυνατότητα από τους τρεις λόγους που αναφέρω και από άλλους βέβαια. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες του καταναλωτή, που είναι περίπλοκες, διότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η δημιουργία καταναλωτικής αξίας που διδασκόμαστε στα πανεπιστήμια είναι κάτι το οποίο δεν πληρεί τα συμφέροντα των καταναλωτών. Ο, ο καταναλωτής αναπτύσσει κάποιες απαιτήσει, αλλά ίσως να μην ίσως δεν ανταποκρίνεται αυτό απόλυτα στην αλήθεια, διότι ο ιδεώδης καταναλωτής είναι αυτός που θα έκανε, ε, θα, θα, ε, είχε τις προσδοκίες αυτές. Τώρα υπάρχει και ένα δεύτερο στοιχείο που είναι η ε, στατική marketing των εταιριών. Και αυτό επηρεάζει και, την, και τις απαιτήσει για την ποιότητα προϊόντων τα οποία θα προχωρήσουν στην μεταποίηση. Και τέλος τα νέα προϊόντα τα οποία έρχονται στην αγορά, διατίθενται στην αγορά και μιλώ για πραγματικά νέα προϊόντα, όχι για τροποποιημένα προϊόντα. Τέλος πάντων, τι μπορούμε να κάνουμε ή τι θα έπρεπε να κάνουμε. Είναι η τρίτη μου αυτή παρατήρηση. Νομίζω ότι ο βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των αγροτών στην αγορά μέσα στα πλαίσια της ε, διατροφικής αλυσίδας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Θα, προτείνω, θα σας προτείνω 7 ε, ενδεχόμενα συμπεράσματα. Μπορούν να προσθεθούν και άλλα στα σχόλια αυτά. Ορισμένα από αυτά περιλαμβάνονται ήδη στο σχέδιο εκθέσεως του κ. Μποβέ. Νομίζω ότι πάντως το πρώτο και πιο περίπλοκο που δεν συζητήθηκε πολύ ευρέως είναι τα κινήματα καταναλωτών. Όσοι είστε οικονομολόγοι εδώ και νομίζω ότι θα είστε το λιγότερο καμιά δωδεκαριά, το ίδιο ε, αν ζητήσω δηλαδή να σηκώσω τα χέρια τους οι δικηγόροι, άλλοι, θα, άλλοι δώδεκα θα σηκώσω τα χέρια και ούτω καθεξής. Αν όμω ρωτήσω πόσοι από εσά είστε καταναλωτέ, τότε θα σηκώσετε όλοι τα χέρια. Παρόλα αυτά, τα κινήματα καταναλωτών συνήθω είναι ασθενή και οι καταναλωτέ είναι συνήθω ανίκανοι να επιβάλλουν τα δικαιώματά του στι αγορέ. Στην Πολωνία διαρωτηθήκαμε γιατί οι καταναλωτές δεν είναι διατεθειμένοι να αγωνιστούν για τα δικαιώματά τους. Και υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις, πάντως η βασική είναι ότι στην ουσία η χαμηλή τιμή μονάδας ενός προϊόντος, ας πούμε λίγα ευρώ ανά κιλό, εάν η ποιότητα του προϊόντος είναι χαμηλή και δεν μας ικανοποιεί, δεν, δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ, γιατί δεν είναι και σημαντική η ζημιά. Πρόκειται για μια αδυναμία του καταναλωτικού κινήματος και είναι διπλά αρνητική. Αφενός διότι οδηγεί σε χαμηλότερο εισόδημα των αγροτών, αλλά και από την άλλη μεριά διότι εμείς καταναλωτές εν τέλει ε, αγοράζουμε τρόφιμα χαμηλότερης ποιότητας. Δεύτερο, η προώθηση άμεσων σχέσεων ε, αγροτών καταναλωτών. Πολλά έχουν λεχθεί σχετικά. Στην ουσία πρόκειται για μια προσπάθεια να καταργηθεί ο μεσάζων. Αυτά έχουν ήδη συζητηθεί. Το τρίτο είναι η ενθάρρυνση της δημιουργίας οργανώσεων αγροτικών παραγωγών. Δεν ξέρω για ποιο λόγο και δεν θα μπορούσα να σας πω για ποιο λόγο φαίνονται απρόθυμοι οι αγρότες να συνεργαστούν μεταξύ τους. Το κατανοώ εν μέρη για τις πρώην σοσιαλιστικέ χώρες, όπου η συνεργασία αυτή ήταν αναγκαστική. Αλλά είναι δύσκολο για μένα να κατανοήσω για ποιο λόγο, παρόλη την χαμηλή τους αγοραστική δύναμη, είναι απρόθυμοι οι αγρότες να ε, συνεργαστούν σε καπιταλιστικές χώρες. Τώρα το τέταρτο, η προώθηση σύντομων, ε, βραχιών δηλαδή, αλυσίδων ε, προμήθεια τροφίμων. Για παράδειγμα, εστιατόρια. Εκεί μπορεί η συντόμευση αυτών των διαδρομών να ε, βοηθήσει πραγματικά. Αυτές είναι soft actions, γιατί δεν απαιτούν παρέμβαση στην ισχύουσα νομοθεσία. Υπάρχουν όμως και άλλες δράσεις που μπορώ να ονομάσω hard actions, τις λέω έτσι εγώ, και που απαιτούν αυτές νομοθετικές παρεμβάσεις και που εν μέρη, όπως είδαμε και στη συζήτηση, μπορούν να γίνουν αποδεκτές και άλλες όχι. Για παράδειγμα, η παρακολούθηση της ε, αγροδιατροφικής αλυσίδας και ορισμένες άλλες παρεμβάσεις, κατάργηση ορισμένων ανεπιθύμητων διαδικασιών και τέλος υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Συμπεραίνοντα, θα πω το εξή. Μπορούν να ληφθούν τέτοιε δράσεις, αλλά αυτές απαιτούν συνένεση όλων των ενδιαφερομένων μερών, αφού απαιτούν σημαντικές νομοθετικές αλλαγές που θα αντιβαίνουν στα συμφέροντα μεγάλων επιχειρήσεων. Μία μεγάλη επιχείρηση, μία από τις 50 μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κόσμο και με έναν προϋπολογισμό μεγαλύτερο από πολλών χωρών, εποφελήθηκε πολύ από την κρίση. Φανταστείτε λοιπόν μια τόσο μεγάλη επιχείρηση τι είδους βαρύτητα έχει ε, στις ε, πολιτικές αποφάσεις. Εν πάση περιπτώσει δράσεις είναι δυνατόν να, να αναλυθούν και εν τέλει θα αποδώσουν σημαντικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ καθηγητά. Τελειώσαμε με όλους τους εμπειρογνώμονες. Έχουμε ακόμη μερικά λεπτά για να μιλήσουμε και να αφήσουμε στο τέλος το λόγο στον Ζωζέ Μποβέ για να τελειώνει. Ο κύριος Χάρκιν. Μετά ο κύριος Ντόρφμαν. Κυρία Άρκιν, συγγνώμη. Ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους ε, όσους πήραν το λόγο και έκαναν παρουσία σήμερα το απόγευμα και ευχαριστώ και τον κύριο Μποβέ. Πολλά από τα θέματα αυτά καλύφθηκαν και θα προσπαθήσω να αναφερθώ σε πράγματα που υπόθηκαν. Κάτι από αυτά που υπόθηκε σήμερα είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την υφιστάμενη νομοθεσία και τα εργαλεία που έχουμε. Νομίζω ότι έχει νόημα που το λέτε αυτό, αλλά πρέπει να δούμε ορισμένα, όπως πριν τόσο χάρη την οδηγία για τις αθέμητες συμπορικέ πρακτικές όταν ε, θα ε, έχουμε να κάνουμε με την παραπλανητική διαφήμιση. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις προς τους καταναλωτές και επίσης θα πρέπει να δούμε ε, και την οδηγία για τις χρηματοπιστωτικές αγορές και νομίζω ότι έτσι θα αυξήσουμε όλη τη διαφάνεια στις αγορές παραγόγων και αυτό θα μας βοηθούσε να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει μικρότερη αστάθεια στις τιμές. Σίγουρα είδαμε υπερβολική ασταθή στις τιμές στο παρελθόν και νομίζω ότι αν είχαμε παράγωγα δυνάμει αυτή τη συγκεκριμένη οδηγία, ε, καθώς ε, υπάρχει κάποια αποπτία και διαφάνεια στις ΗΠΑ, αλλά δεν υπάρχει εδώ, αν μπορούσαμε και εμείς να πετύχουμε κάτι τέτοιο, νομίζω ότι αυτό θα μείωνε της, ε, την αστάθεια των τιμών και θα βελτίωνε τη σταθερότητα στην αγορά. Μπορούμε λοιπόν ε, να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά στο πλαίσιο ε, των δραστηριοτήτων μας αναφερθήκατε στην πολιτική ανταγωνισμού. Αυτή η πολιτική ανταγωνισμού δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα στην αλυσίδα. Επίσης πρέπει να υπάρχει κατάλληλη παρέμβαση και νομίζω ότι ο τελευταίος ε, ομιλητής ε, αναφέρθηκε σε αυτές τις ε, soft και hard δράσεις. Δεν θα αναφερθώ εγώ λεπτομερώς. σα άκουσα τι είπατε. Τώρα για τα τελευταία δύο σχόλια που θέλω να κάνω και πάλι αναφερθήκατε στους ε, κυρίαρχους συνδεσμούς ε, στην στη διατροφική λύσιδα και πρέπει να δούμε τι έχει γίνει σήμερα ο αυτός ο δεσπόζων σύνδεσμος ε, και ίσως πρέπει να δούμε πώς ακριβώς μπορούμε να εφοδιάσουμε τη διατροφική αλυσίδα όμως η παραγωγή ποτέ δεν ήταν αυτός ο δεσπόζων κρίκος και νομίζω ότι φάνηκε με σαφήνεια ότι αν δούμε ε, το ότι είχαμε αύξηση ε, της αξίας και του εισοδήματος σε όλους τους τομείς από το 1995 στο 2005, αλλά δεν είδαμε αύξηση στο εισόδημα των παραγωγών. Επίσης, ακούμε ότι θα πρέπει η Γεωργία να είναι βιώσιμη και προσανατολισμένη στην αγορά, δηλαδή θα πρέπει να λαμβάνουν και ένα λογικό εισόδημα οι Γεωργοί για την εργασία τους. Και ε, είπαν ε, πολλοί ότι ένα μεγάλο ποσοστό της οδημότητας των Γεωργών προέρχεται από τις ε, άμεσες ενισχύσεις. Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Έχουμε λοιπόν κάποιες soft δράσεις και κάποιες hard δράσεις. Θα πρέπει να το επιλύσουμε αυτό το θέμα τώρα έτσι ώστε να μπορέσουμε ε, το 2013 να αναθεωρήσουμε την κοινή αγροτική πολιτική με έναν βιώσιμο τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Χάρκιν. Ο κύριος Ντόρφμαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν αναζητούμε τώρα καλούς και κακούς μέσα στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρξει ισότιμη μεταχείριση των διαφόρων εταίρων εντός εισαγωγικών. Επανέρχομαι στον πρώτο γύρο της, ε, των συνομιλιών που κάναμε σήμερα το απόγευμα. Για παράδειγμα, η πρόταση να θεσπιστούν δίκαιες τιμές. Ωραία, αλλά ποιες είναι οι δίκαιες τιμές και πώς θα εφαρμοστούν οι δίκαιες τιμές. Άλλωστε το εμπόριο πρέπει να παραμείνει ελεύθερο, έτσι πιστεύω. Κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις πρέπει να σκεφτούμε για την αγροδιατροφική αλυσίδα. Δύο μου φαίνονται σημαντικές. Και με αυτές συνδυάζω και μια ερώτηση προς τον εκπρόσωπο της Eurocommerce. Πρώτα το θέμα των στόχων των πληρωμών. Αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα για την γεωργία και για το συνεταιριστικό κίνημα των αγροτικών παραγωγών. Εάν συμφωνήσουν οι αλυσίδες ε, υπερκαταστημάτων με ένα ανώτατο όριο πληρωμών, δεν θα τίθεται πλέον θέμα ανταγωνισμού. Άρα θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία για κάτι τέτοιο. Κάτι που μου φαίνεται σημαντικό είναι ότι δεν είναι δυνατόν εκ των υστέρων να επιβάλλονται τροποποιήσεις των συμβάσεων. Ενώ σημειώνεται, σημειώνονται τέτοια φαινόμενα. Και αυτό προκαλεί σημαντικά προβλήματα στην αγορά των αγροτικών προϊόντων. Ένα τελευταίο είναι το θέμα της ρύθμισης το θέμα της αυτορύθμισης για κατάλοιπα φυτοφαρμάκων. Έχει σημειωθεί το φαινόμενο τελευταία αλυσίδες υπερκαταστημάτων να έχουν θεσπίσει των εισαγωγικών δικούς τους κανόνες για, ε, τα, περιεχόμενα, για, για τα περιεχόμενα τέτοιων καταλήπων. Κάτι το οποίο στερεί οποιαδήποτε αξιοπιστία από τις ρυθμίσεις αυτές που δεν βασίζονται σε, ε, σε επιστημονική θεμελίωση, ούτε μπορεί να πει κανένα ότι μια λυσίδα υπερκαταστημάτων είναι καλύτερη από μια άλλη και αυτό στα μάτια του καταναλωτού μπορεί να μην καταλαβαίνει τέτοια πράγματα, ούτε μπορεί να γνωρίζει ε, τι είναι προτιμότερο να υπάρχει ε, λίγο κατάλοιπο από το τάδε προϊόν υγειονομική προστασίας και περισσότερο από άλλο ή το αντίθετο δεν μπορεί να τα γνωρίζει αυτά. Εδώ χρειάζεται κάποια παρέμβαση και νομίζω ότι αποτελεί νομοθετικό καθήκον να πάυσει αυτή η αταξία και μου φαίνεται αρκετά παράλογο το ότι καθένας μπορεί να θεσπίζει κανόνες ιδιωτικούς για την υπόθεση αυτή. Η κυρία Μορβάη. Πολύ ενδιαφέρουσα η σημερινή συζήτηση. Ακούσαμε τοποθετήσεις ε, για ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό δηλαδή το δίκαιο εισόδημα για τους αγρότες. Όμως ε, μιλάμε εδώ για τους Ευρωπαίους αγρότες ε, και όχι για αγρότες που βρίσκονται σε συγκεκριμένη κατάσταση, δηλαδή σε χώρες μετακομμουνιστικού καθεστώτος ε, εδώ. Μιλήσαμε και για θέματα ανταγωνιστικότητα. Η ανταγωνιστικότητα είναι μία από τι κύριε έννοιε. Θα πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμό. Όμω, πώ θα διασφαλίσουμε τον ανταγωνισμό, κυρίω αν μιλάμε για μικρού παραγωγού. Αν, παραδείγματο χάρη, οι αγρότε αυτέ θα πρέπει να ανταγωνιστούν με πάρα πολύ μεγάλε βιομηχανικέ εκμεταλλεύσει. Και αν προσπαθήσουμε να υπάρξει ε, τελικά μια διαφορετική ανάπτυξη. Δηλαδή είδαμε ότι σε κάποιες χώρες στο παρελθόν υπήρξε εθνικοποίηση κάποιων μεγάλων επιχειρήσεων. Όμως ε, εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, την ε, πραγματικότητα της αγοράς και να σας πω πού είναι το δίκαιο εισόδημα στην κατάσταση αυτή θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το σημείο αφετηρίας, δηλαδή ήδη βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί σε μειονεκτική θέση. Στην Ουγγαρία είχαμε το 25% ε, του πληθυσμού είναι γεωργοί και σήμερα δυστυχώς δεν λαμβάνουμε ένα ποσοστό σε πληρωμές που να καλύπτει τη γεωργική δραστηριότητα. Και πώς μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί αυτή οι παραγωγή. Εμείς θέλαμε να προωθήσουμε κάποιες ε, τροπολογίες ε, στην έκθεση για να είμαστε σίγουροι για το ότι μιλάμε για τη βιωσιμότητα και τον ανταγωνισμό. Υπάρχει μια πολύ σημαντική μελέτη στην Ουγγαρία, την έχουμε δώσει στον συγητή και θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε για την εξαιρετική δουλειά του. Honorable Rubins. Rubins. Και μετά Νικολέσκου. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Μποβέ, όπως και τους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι πήραν το λόγο σήμερα, διότι αυτή η ακροασία ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ χρήσιμη. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στο θέμα της συζήτησής μας σήμερα, δηλαδή για, μια, για την άσκηση μιας σωστής αγροτικής πολιτικής. Θα έπρεπε λοιπόν να ληφθούν μέτρα που θα απαγορεύουν στη μεγάλη διανομή, στα δίκτυα μεγάλης διανομής, να αγοράζουν τα προϊόντα των παραγωγών σε χαμηλότατες τιμές, προϊόντα μη συσκευασμένα που συσκευάζουν τα ίδια τα σούπερ μάρκετ και τα πολλούν ως προϊόντα δικά τους. Εγώ έρχομαι από τη Λετωνία, παίρνω το αεροπλάνο πολύ συχνά και στο αεροπλάνο μου δίνουν ζάχαρη. Ζάχαρη συσκευασμένη σε ένα χάρτινο σακουλάκι, το οποίο απλώς φέρει το όνομα της εταιρείας. Δεν υπάρχει κανένα, καμία ένδειξη από πού έρχεται αυτή η ζάχαρη, ποιος την έχει παράγει. Θα έπρεπε λοιπόν αυτά να τα ρυθμίσουμε. Εγώ θεωρώ ότι η αδικία που πλήττει τους γιοργούς μας βρίσκεται στις δικές μας πρακτικές και θέλω να σταθώ σε αυτά τα οποία είπε η Ουγγαρέζα συνάδελφος με την οποία θέλω να συμφωνήσω. Μα για ποια δικαιοσύνη μιλάμε όταν ένας εσθονός Γιοργος κερδίζει τέσσερις φορές λιγότερο για το ίδιο προϊόν από ότι η γεωργοί της παλαιάς Ευρώπης. Για όταν μιλάμε για την Ευρώπη 2013-2020 και τη γεωργία της, ελπίζουμε πολλά, και, αλλά δεν αυξάνουμε με τίποτα τον προϋπολογισμό. Και οι εμπειρογνώμονες λένε, μα πώς θα τον εξισορροπήσετε τούτον τον προϋπολογισμό, αν τα παλιά κράτη-μέλη δεν απαρνηθούν τις επιδοτήσεις τους. Αυτά είναι θέματα τα οποία είναι ανοιχτά, για τα οποία δεν έχουν βρεθεί απαντήσεις. Και θεωρώ ότι αν εργαστούμε επί του κειμένου του κυρίου Μπόβε θα τη βρούμε τη λύση. Ευχαριστώ κύριε Ρούμπινς. Ο κύριος Νικουλέσκου, αντιπρόεδρος, έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ, πρόεδρε. Όλες οι ιδέες του κυρίου Μποβέ είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αλλά δεν πρέπει να χάνουμε την ουσία από μπροστά μας. Και κυρίως μη χάνουμε τον ορίζοντα. Εγώ έρχομαι από πω την Ρουμανία, χώρα που τελευταία πολύ συζητήσαμε το θέμα του ποσού που πληρώνονται και ένας εθνικός βουλευτής πρότεινε να κλείνουν τα σούπερ μάρκετ την Κυριακή. Αυτό είναι κακό πράγμα, διότι ε, ε, ε, δεν είναι σωστό. Η, λύση λοιπόν δεν είναι να κλείνουμε μαγαζιά ή οτιδήποτε άλλο, είναι να αυξάνουμε την ανταγωνιστικότητα, συνεταιρισμοί, εξυγχρονισμός των μονάδων, και να διευκολύνουμε την είσοδο των γεωργών στο εμπορικό κύκλωμα. Αυτά. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστώ Νικουλέσκου. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους εμπειρογνώμονες και όλα όσα μας είπαν. Δύο πράγματα και μετά θα δώσω το λόγο στον Ζωζέ για να κλείνει. Πρώτα απ' όλα, ε, κατάθεση τροπολογιών 18 Μαΐου στις 12 τελική προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών στην έκθεση ΒΟΒΕ. Θα τα εγκρίνουμε όλα αυτά στις 28 Ιουνίου για να πάνε στην Ολομέλεια το Σεπτέμβριο. Θυμίζω επιπλέον και πιο συγκεκριμένα στο Ζωζέ, συγχαίροντας για την εξαιρετική δουλειά, ότι το φθινόπωρο θα έχουμε τρία μέτρα, νομοθετικά μέτρα για την ποιότητα, έκθεση σκοτά, θα έχουμε την έκθεση για τις προβληματικές περιοχές και θα έχουμε, και μας το είπε Επίτροπος ε, πριν από δύο εβδομάδες στο Στρασβούργο, ένα πακέτο μέτρων για τη διαχείριση της αγοράς που θα παρουσιαστεί μετά από τη λήξη των εργασιών της ομάδας υψηλού επίπεδου. Τρία σημαντικά νομοθετικά μέτρα στα οποία θα μπορούσαν να ενσωματωθούν και ορισμένες από τις προτάσεις που άκουσα σήμερα. Παρακαλώ λοιπόν τους συναδέλφους να προσέξουν όλες αυτές, όλα αυτά τα θεσμικά ραντεβού που έχουμε, θα έχουμε το φθινόπωρο ώστε να θησαυρίσουν όλα όσα ακούσαν εδώ μέσα. Ζωζέ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα προσπαθήσω να ολοκληρώνω με λίγα λόγια γιατί όλοι είναι κουρασμένοι. Ε, είχαμε πολλές συζητήσεις, δεν θα μακρηγορήσω. Ε, εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που ήρθαν, όλους τους εμπειρογνώμων. όλοι που εκπροσώπησαν τη διανομή, τα πανεπιστήμια, τα πανεπιστήμια και τα Ηνωμένα Έθνη και φυσικά την ΟΚΕ. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν για τη δουλειά σας, για τη συνεισφορά σας που επέτρεψε στους βουλευτές να καταλάβουν καλά την πολυπλοκότητα του πράγματος και ότι δεν μπορεί κανείς να είναι απλοϊκός και αφελής αυτού του είδους τις συζητήσεις. Υπάρχουν προβλήματα ρυθμιστικά, νομοθετικά και πίσω από όλα αυτά υπάρχει και πολιτική φυσικά. Το πολιτικό όραμα. Αυτό το οποίο ανέφερε και ο συνάδελφος Καπουλασάντος. Είναι φανερό ότι δεν μπορούμε εμείς να εξετάζουμε αυτά τα ζητήματα χωρίς να θέτουμε το πολιτικό πρόβλημα. Και επανερχόμαστε έτσι στο 1957 στη συνθήκη της Ρώμης και τη δημιουργία της ΚΑΠ. Τρεις στόχοι. Ανεφοδιασμός, ποσοτικός αφοδιασμός των Ευρωπαίων πολιτών, σταθερότητα των τιμών και τρίτο οι χώροι εκεί να έχουν ένα εισόδημα αντίστοιχο με τις άλλες κοινωνικές κατηγορίες το το τρίτο κεφάλαιο το ξεχνούσαν συνεχώς τις κοινέ αγροτικές πολιτικές και είναι φανερό ότι αυτή η έκθεση επανεντάσσεται στην εξισορρόπηση αυτής της πολιτικής. Εάν δεν το κάνουμε τότε όλη αυτή η σπήρα ε, με ψιλογιώτα φυγής από τη Γεωργία θα συνεχίσει η προστασία των θέσεων απασχόληση είναι 12 εκατομμύρια θέσεις αγροτών, χωρικών. Το να τους αγνοήσουμε θα ήταν αυτοκτονία για την Ευρώπη, κοινωνική, οικονομική, αλλά και ε, τροφιμικής επισητιστικής κυριαρχίας. Δύο ζητήματα. Ή ο χωρικός αμείβεται σύμφωνα με την εργασία του ή με τη συνεισφορά των συμπολιτών του των Ευρωπαίων μέσω της φορολογίας. Δηλαδή από τη μια πουλάει τα προϊόντα του και από την άλλη ενισχύεται μέσα από τους φόρους που πληρώνουν οι συμπολίτε του. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένας γεωργός, νέος γεωργός που να θέλει να εγκατασταθεί, να ξεκινήσει δηλαδή και να ζει με τις επιδοτήσεις. Θέλει ένας νέος παραγωγός να δουλέψει, να βγει στην αγορά και να δουλέψει από την παραγωγή του και από τη δουλειά του. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτές οι άμεσες ενισχύσεις έτσι όπως διανέμονται είναι άνισες, αλλά δημιουργούν και τέτοιου είδους σχέσεις εισοδηματικές που είναι και που είναι αντικονομικές. Αν εμείς θέλουμε μία πολιτική που βασίζεται στη σωστή αμοιβή συνδεδεμένη με το κόστος παραγωγής, τότε έχουμε μια οικονομία δυναμική που επιτρέπει και μια ισορροπία μεταξύ παραγωγών. Πολλοί το έπανε ότι θα πρέπει να έχουμε και μια κυραγώγηση, της, ε, έναν έλεγχο της παραγωγής για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τις τιμές. Όταν βλέπουμε εμείς ότι οι κοινέ οργανώσεις αγοράς έχουν απογυμνωθεί αλλά επέτρεπαν όμως το παρελθόν να οργανώνουν τα διάφορου τους διάφορους ε, τομείς και εκτός από το μαλακό στάρι όλα, όλες οι υπόλοιπες κόες ήταν ρυθμισμένες. Πώς τα κράτη λοιπόν επέτρεψαν κάτι τέτοιο, δηλαδή την εξασθένιση των, της κοινής, των κοινών οργανώσεων αγοράς χωρίς να έχουν εναλλακτικά μέσα στη διάθεσή τους. Πρέπει να είμαστε λοιπόν ρεαλιστές και να μην χάνουμε και τον πολιτικό μας ορίζοντα. Γι' αυτό αυτή η συζήτηση είναι εγκάρσια. Εγώ νομίζω ότι σήμερα έχουμε τα μέσα να προχωρήσουμε και αυτό που θέλω να πω είναι ότι χάρηκα πολύ με τις τοποθετήσεις των βουλευτών και ελπίζω ότι για τις τροπολογίες μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμη πιο μακριά από τι προτάσεις μου. Αυτό εύχομαι εγώ στο κείμενό μου, δηλαδή να το σκληρύνουν το κείμενο οι βουλευτές. Και χθε εγώ πήρα ένα σημείωμα για την έκθεσή μου από τις γαλλικές αρχές που λένε ότι είναι καλή έκθεσή μου, αλλά μπορούσαμε να το τραβήξουμε πιο μακριά σε ορισμένους τομείς. Ε, λοιπόν, εγώ το λέω στους βουλευτές, Γιούρια, διότι στα πλαίσια των τροπολογιών μπορούμε να λύσουμε τα πράγματα. και το, όταν ε, το συζητήσαμε βέβαια και σήμερα το πρωί με τους, ε, με τους υπεύθυνους των ομάδων για να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις τροπολογίες και να είναι αποτελεσματική έκθεση. Εύχομαι πάντως να συνεργαστούμε. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργατικότητά σας και ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν από μακριά για να παρακολουθήσουν αυτή τη συζήτηση και που θα μπορέσουν και αυτοί να εμπλουτίσουν με τη συνεισφορά τους διότι χρειαζόμαστε εμείς οργανώσεις της αγροτιάς, της κοινωνίας των πολιτών, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μία δίκαιη ΚΑΠ. Ευχαριστώ. Σίγουρα, σίγουρα. Συλλογική προσπάθεια θα καταβάλουμε. Τελειώνουμε. Επόμενη συνεδρίαση 10 Μαΐου με την Ισπανική Προεδρία θα συναντηθούμε και θα συζητήσουμε για την αντιγωνιστικότητα στη Γεωργία.